Αγαπητοί συνάδελφοι, λέω να αρχίσουμε. Θα είδατε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση να την εγκρίνουμε. Σας πληροφορώ ότι σύμφωνα με αυτά που είχαμε αποφασίσει στην προηγούμενή μας συνεδρίαση, το σημείο για τις αγορές κτηρίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητηθεί παρουσία του Γενικού Γραμματέα Κλάους Βέλε στις 3 και μισή. Θα αρχίσουμε λοιπόν, θα σταματήσουμε στις 3.30 μέχρι τις 4 και 4 για να ακούσουμε το Γενικό Γραμματέα και την εισηγήτριά μας την Μόνικα. και μετά θα δούμε και τι ερωτήματα μπορεί να τίθενται ή να τεθούν στο Γενικό Γραμματέα μετά από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάναμε με τον Αντιπρόεδρο Βιδάλ Κουάδρα στην περασμένη εβδομάδα. Μετά είπαμε να γίνουν ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τις 5 και 4 με 5 και 20 μέχρι τις 6 και στις 16.30, στις 18.30 κανονικά θα τελειώσουμε. Εγκρίνεται η μέρες διάταξη, εγκρίνεται. Ανακοινώσεις θα έχει η τα νέα της Κομπούς. Αν δεν υπάρξουν σχόλια ή αντιρρήσεις και για τα πρακτικά της 7ης Νοεμβρίου θα εγκριθούν και αυτά. Τώρα, να πως να αρχίσουμε, τι λέει ο Γιάνν Λουκ και η Άννα. Το πρωί συναντηθήκαμε με μια αντιπροσωπεία του τρίου προεδριών για τους νέους ιδίους πόρους μέσα στα πλαίσια της κέντρου δημοσιονομικών προοπτικών του ε, επομένου έτους. Η συνάντηση αυτή ήταν σύντομη και ίσως να σας πω πολύ γρήγορα τι έγινε στα 4, 5 και 6 δηλαδή. Και οι δύο εισηγητές, Ζανλούκ Ντεάν και Άννα Γένσεν, να μας πούν τι έγινε σε αυτή τη σύντομη. Θέλετε να τα πω εγώ? Α, ε, θα τα πω εγώ λοιπόν. Λοιπόν, έχω το λόγο. Με την έγκριση των εισηγητών και εισηγητριών. Λοιπόν, καταφέραμε όλες οι διαπραγματεύσεις του επόμενου πολιετούς διαπραγματευτικού πλαισίου για τις, ε, να γίνουν παράλληλα μέσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Παράλληλα, Κοινοβούλιο-Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, στο ειδικό του επίπεδο δηλαδή, σε επίπεδο υπουργών και αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, θα, κάνει, θα συζητήσει το θέμα των δημοσιονομικών προοπτικών και μετά θα στραφεί σε εμά. Θα μας πει ορίστε η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, τώρα μπορείτε να τη δεχτείτε ή να την απορρίψετε ή να κάνετε τροποποιήσεις. Αυτή η διαδικασία βέβαια μας έβαζε σε πολύ δύσκολη θέση. Στο εξή από την πρώτη μέρα θα ε, παίζουμε κάποιο ρόλο. Δηλαδή γίνανε τρεις συναντήσεις ανταλλαγών απόψεων προς το παρόν γιατί και το ίδιο το Συμβούλιο δεν μπορεί να αρχίσει ακόμα τη διαπραγμάτευση. Οι εθνικές αντιπροσωπείες δεν έχουν την δέουσα εντολή. Στις 12 Σεπτεμβρίου έγινε η πρώτη τέτοια συνάντηση για τα γενικά, για τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών, για την κατανομή ανακατηγορία. Δεύτερη συνάντηση έγινε το Νοέμβριο για τις προτάσεις της Κομισιόν ως προς την ΚΑΠ και την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής. Οι αυτές ήταν οι δύο μεγάλες κατηγορίες, η Α και Β καθώς και δύο. Και το πρωί σήμερα έγινε μια ανταλλαγή απόψεων, η τρίτη, για τους νέους ιδίους πόρους. Στην ουσία, μονόλογος ήταν εκ μέρους του Κοινοβουλίου προς τους τρεις Υπουργούς Εξωτερικών. Προτείναμε λοιπόν και καταφέραμε να εκπροσωπηθεί και η Κομισιόν, Επίτροπος Λεβαντόσκη. Προτείναμε πρώτον για το Κοινοβούλιο πολιτική συμφωνία για τους νέους για τους νέους ιδίους πόρους να είναι όρος για την έγκριση του πολιετούς σχεδίου. Δεν συμφωνεί δηλαδή το Κοινοβούλιο για όλες τις δαπάνες και την αναθεώρησή τους. Δεύτερο μήνυμα, τρία μηνύματα είχαμε πει. Δεύτερον, αυτά που είχαμε πει και στην Κομπού την περασμένη εβδομάδα με βάση τις προτάσεις των εισηγητών και εισηγητριών. Δηλαδή ότι θεωρούμε ότι οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την Κομισιόν είναι μια σωστή βάση συζήτησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τις δεχόμαστε 100% ούτε ότι δεν επιφυλασσόμεθα να προτείνουμε και κάτι καινούργιο. αλλά θεωρούμε ότι είναι μια βάση επί της οποίας μπορούμε να συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Θα δούμε αν στη συνέχεια χρειαστεί ή όχι να διευρυνθεί αυτή συζήτηση. Θεωρούμε πάντως είναι μια καλή βάση. Και επίσης επέμεινα ότι ότι λέγω η, το πνεύμα του Κοινοβουλίου από την αρχή για τους ιδίους πόρους είναι να μην τροποποιηθεί η συνθήκη. Εμείς δουλεύουμε με βάση την ισχύουσα συνθήκη. Δεν ζητούμε νέες δικαιοδοσίες ούτε για την Ένωση ούτε για μας ζητούμε την εφαρμογή των συνθήκων που προβλέπουν ήδη τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ιδιών πόρων. εφόσον βέβαια εγκριθούν ομόφωνα από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και αυτό είναι όπως βλέπετε θέμα συνομοθεσίας όπου το Κοινοβούλιο δεν περιορίζεται στο να εκφράσει μια γνωμοδότηση. Επ' αυτού όμως το Κοινοβούλιο προς στιγμή δεν ζητάει τροποποίηση των συνθήκων. Αυτό ήταν καλό να το τονίσουμε γιατί ακούγεται από εδώ και από εκεί και στις Βρυξέλλες και αλλού ότι ζητάμε λέει νέα συνθήκη. Εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να δηλώσουμε ότι για αυτό το θέμα των ιδίων πόρων είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και νομικώς μετριόφρονες. Είμαστε φιλόδοξοι ως προς το στόχο, αλλά ως προς τα νομικά μέσα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε είμαστε πολύ μετριόφρονες. Να χρησιμοποιήσουμε την ισχύουσα συνθήκη. Χωρίς να αμφισβητήσουμε και αποφάσεις που έχουν ίδια ισχύ με τις συνθήκες όπως το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων. Αυτά. Λοιπόν, μήπως οι εισηγητές θέλουν να προσθέσουν τίποτα. Ο Ιωάννης Λουκάς, η Άννα. Μόριστε Άννα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Δανική Προεδρία έχει πει ότι σχεδιάζει να συνεχιστούν οι συζητήσεις με έξι συναντήσεις και από ό,τι λένε, μάλλον θα μπορέσουν να, να πετύχουν να υπάρξει συνένεση σε αρκετά σημαντικά σημεία. Έτσι, τον Ιούλιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι δυνατόν να γίνει ε, δεκτή μία δέσμη αρχών, ε, όχι συγκεκριμένων αριθμητικών στοιχείων, αρχών. Και ο φάκελος αυτός θα διαπιβαστεί στον κύριο Φων Πάι και τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν για τα νούμερα σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές και Ελπίζουμε μέχρι τον Οκτώβριο να έχει επιτευχθεί μια συμφωνία. Μία διπλή διαδικασία προβλέπουν, δηλαδή να γίνει μια συζήτηση για τη βασική νομοθεσία και την μεταρρύθμιση κοινή γεωργική πολιτικής, διαρθρωτικών ε, προγραμμάτων, ερευνητικών προγραμμάτων και ούτω καθεξής. Τα νομικά κείμενα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν στο Συμβούλιο και παράλληλα θα γίνονται και οι συζητήσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Οι συζητήσεις δηλαδή για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα γίνονται εκ παραλλήλου. Και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό. Γιατί εάν οι χώρες μπουν στη διαδικασία να ότι θα πληρώνουν τόσο και όχι παραπάνω και κάποιες άλλες χώρες ε, ζητούν χρηματοδότηση, εκεί θα υπάρχουν δυσκολίες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο έχετε στο φάκελό σας είναι ένα έργα, έγγραφο εργασίας από τον κύριο Ντεάν και την υποφαινομένη που σας δίνει κάποια στοιχεία για τους ίδιους πόρους ε, που έχουμε καταλήξει μέχρι τώρα με το Συμβούλιο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διάγραμμα που δείχνει ποιες προτάσεις είναι επιτάπητος συμπεριλαμβάνονται και το θέμα των νέων ίδιων πόρων, η πρόταση για τον ΦΠΑ, η πρόταση για αυτοφόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δηλαδή νομίζω ότι έτσι είναι πιο εύκολο να δείτε όλοι τι προτάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι μέχρι στιγμής. Είναι το έγγραφο εργασίας παριθμών 1 αυτό. Νομίζω ότι μπορείτε έτσι γρήγορα γρήγορα να έχετε μια ιδέα με τις ε, συνοπτικές αυτές ε, προτάσεις. Κατά την άποψή μου αλλά και του κυρίου Ντεάν θα συνεχιστεί η επεξεργασία των προτάσεων αυτών. Εμείς βέβαια επιφυλασσόμεθα, γιατί μπορεί να πέσουν και άλλε προτάσει στο τραπέζι. Έχουμε όμω την πρόταση για το ΦΠΑ και το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που είναι και η βάση των συζητήσεων για, νέους, για του νέου ίδιου πόρου. Ο φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τέλο πάντων η πρόταση για ένα τέτοιο φόρο, συζητείται στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή οίκων, την Οικονομική Επιτροπή. Στο Συμβούλιο το Νοέμβριο στο ΕΚΟΦΗΝ συζητήθηκε η πρόταση αυτή για το φόρο χρηματοπιστωτικό συναλλαγών. Ήταν μια αρχική συζήτηση, αλλά ακόμη δεν έχουμε σχηματίσει μια εικόνα με βάση τις συζητήσεις αυτές για το ποια ήταν η έκβαση. Είναι η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά, την Αρμόνιση. Ε, εκεί αποφασίζεται, συζητείται ε, ο φόρος αυτός. Και εμείς θα πρέπει να δούμε εν συνεχεία πώς θα λειτουργήσει αυτός ο φόρος ε, ως ε, ένα τμήμα των ιδιών πόρων. Να δούμε τι αρχές θα ισχύουν. Γιατί είναι το θέμα του κατά πόσο ο φόρος αυτός είναι δίκαιος, είναι αναδιαμητικός, αν είναι σταθερός. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να μετρήσουν ενδεχομένω το κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να εισαχθεί αυτός ο νέος φόρος ως ένας νέος ίδιος πόρος είναι αξιόπιστος, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτά είναι τα ερωτήματα μεταξύ άλλων. Αυτά είναι και όσα θα θέλαμε ίσως να πούμε στο Συμβούλιο. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά ε, μιλάμε για μια εισαγωγική φάση ε, στο επίπεδο του Συμβουλίου για τη συζήτηση των ιδιών πόρων. Το έγγραφο εργασία είναι το πρώτο βήμα για να δούμε πώ μπορούμε και εμεί να εργαστούμε στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν ο κύριος Άρτον ε, έχει ζητήσει το λόγο. Voorzitter, dank u wel. Het is een interessant stuk. Ehm, Πρόεδρε, πρόκειται για ένα ενδιαφέρον έγγραφο. Οι Δανείοι και οι Κύπροι είναι πάρα πολύ θαραλέοι άνθρωποι, αλλά την επόμενη χρονιά δεν θα ήθελα που δεν είναι να είμαι στη θέση τους διότι πρόκειται να λάβουν χώρα διαπραγματεύσεις ε, για το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, ε, η αναθεώρηση του προγράμματος ITER και αυτά απαιτούν την ομοφωνία στο Συμβούλιο. Πριν από λίγο απευθύνθηκα στην Κομισιόν και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό και οι δύο ε, μου είπαν ότι για το θέμα αυτό απαιτείται ομοφωνία. Αναφέρομαι βέβαια στους ίδιους πόρους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διερωτώ λοιπόν κατά πόσον ε, προβλέπουμε σωστό χρονοδιάγραμμα, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ολλανδοί ανέκαθεν ήταν κατά του συστήματος των ιδίων πόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για το Υπουργικό Συμβούλιο της Ολλανδίας, αλλά και για την αντιπολίτευση. Εμείς στο σύνολό είμαστε κατά του συστήματος των ιδίων πόρων. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Αυτό το θέμα πρέπει να το θίξουμε σήμερα γιατί η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αυτό και κάνουμε σήμερα, το έκαναμε και τις δύο προηγούμενες φορές και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και του χρόνου. Η Αν Γένσεν μας υπενθύμισε και το χρονοδιάγραμμα της Δανικής Προεδρίας. Τώρα, το γεγονός ότι υπάρχουν ε, έντονες αντιρρήσεις ε, στο Συμβούλιο σε αυτή τη φάση είναι φυσιολογικό, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Σε διαπραγματεύσεις ε, βρίσκονται. Και στην αρχή μάλιστα των διαπραγματεύσεων κάποιοι τότε λένε ότι είναι υπέρ κατά τη τάδε ή τη δίνα λύση. Το σημαντικό είναι να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η ίδια η διαπραγμάτευση. Αν δηλαδή ένα κράτο μέλο ε, θέσει υπό αμφισβήτηση τη διαπραγματεύση, εκεί θα ε, δημιουργηθούν προβλήματα. Δεν ισχύει όμω κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι στο γενικό πλαίσιο που ζούμε και σήμερα, δεν είναι προ το συμφέρον κανενό κράτου να μπλοκάρει τη δρομολόγηση των διαπραγματεύσεων για το μέλλον τη Ένωση. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ούτω ή άλλω Γίνονται, όπω είπα, αυτέ οι διαπραγματεύσει, έχουν ξεκινήσει. Φυσικά, το σημερινό Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ήταν αφιερωμένο κυρίω στην προπαρασκευή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 9η Δεκεμβρίου, στα τέλη δηλαδή τη εβδομάδα. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για του ίδιου ε, πόρου, αλλά μάλλον σε πολύ, πάρα πολύ σύντομη θα ήταν αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Όπω είπε η Ιάν, η αλήθεια είναι ότι οι πραγματικέ διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόνο Επιδάνική προεδρίας, στους προσεχείς μήνες δηλαδή. Το, ε, τώρα πότε θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις δεν το γνωρίζουμε, δεν έχουμε ιδέα. Το χρονοδιάγραμμα, το οποίο όλοι μας εργαζόμαστε προς το παρόν τουλάχιστον, είναι η κατάρτιση ενός εγγράφου τον Ιούνιο από τη Δανική Προεδρία, το οποίο θα κάνει έναν απολογισμό για τις απόψεις των ΜΕΝ και των ΔΕΣ ότι αφορά τα σημαντικά σημεία της συζήτησης και εντό Συμβουλίου και μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και από εκεί και πέρα το Συμβούλιο θα κρίνει από πλευρά του κατά πόσον θα συνεχίσει να εργάζεται σε επίπεδο Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή εάν θα περάσει απευθεία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα που θα πρέπει να το σκεφτούμε και να προετοιμαστούμε αναλόγως. Δηλαδή, πώς θα συνεχίσουμε εμείς τη δική μας ανταλλαγή όταν το ζήτημα πλέον πάει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμη. Θέλω να ευχαριστήσω πάντω του εισηγητέ ε, για αυτό το έγγραφο εργασία. Το είχαν ζητήσει πολλέ πολιτικέ ομάδε και χρειαζόμασταν πράγματι ένα τέτοιο έγγραφο για να δούμε πιο ξεκάθαρα τις διάφορες ε, θέσεις και προτάσει και τι πρακτικέ επιπτώσει, ιδίω για καθένα κράτο μέλο, τις επιπτώσεις που θα έχουν οι προτάσεις ε, που υπέβαλε η Κομισιόν, θα θυμάστε ότι η διάσκεψη των Προέδρων είχε αποφασίσει, αποφάσισε να συγκροτήσει μια ομάδα επαφής, ένα contact group που θα συνεδριάζει περιοδικά για να εξετάζει την κατάσταση και θα προεδρεύει αυτή τη ομάδα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος Μπούζεκ ενημερώθηκα ότι σκεφτόταν να, να συνεδριάσει για πρώτη φορά αυτή η ομάδα επαφής με αυτόν ως πρόεδρο την προσεχή εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ίσως την Τρίτη, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι. Θα σας δώσω τις ε, λεπτομέρειες όταν και εφόσον ενημερωθώ και εγώ σχετικά. Και με τον πρόεδρο Μπούζεκ, αλλά κυρίως και με τον διάδοχό του θα έλεγα, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελική σύνθεση και ποιος θα είναι και ο τρόπος και ο ρυθμός εργασίας αυτής της ομάδας επαφής. Αυτά από μέρους μου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Αν όχι μπορούμε να κλείσουμε τα σημεία 4, 5 και 6 Ο Γενικό Γραμματέα Κλάους Βέλε μόλις έφτασε, τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Ήταν διαθέσιμο και την προηγούμενη φορά, αλλά δυστυχώς εμείς δεν είχαμε χρόνο, γιατί ήταν ο αντιπρόεδρο Βιδάλ Κουάδρα, ε, τον οποίο είχαμε στην ε, επιτροπή μας. Ε, η Μόνικα Χολμάγερ δεν ξέρω αν είναι εδώ. Να μας πει κάποιος αν φτάνει, ναι, που ναι, ναι. βρίσκεται γιατί θα είχα τύψεις. Δεν θα ήθελα να θέσουμε το θέμα αυτό και να το συστήσουμε χωρίς να είναι εδώ η Μόνικα. Α, έφτασε. Και έρχεται και με τους φακέλους της παρέα. Ωραία, μπράβο. Εντάξει, με την ησυχία σου Μόνικα, κάθισε, βολέψου. το λέω κυρίως για το Γενικό Γραμματέα τώρα, στην προηγούμενη συνεδρίασή μας είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την αγορά δύο κτηρίων, σχέδιο το οποίο συζητήθηκε στη διάσκεψη των Προέδρων, μόνο του Αγιέ στι Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο, δεύτερο κτίριο. Πρόσφατα, αποφασι... Ε, μάλλον μάθαμε ότι υπήρχε και ένα άλλο σχέδιο, ένα άλλο πρόγραμμα που εξέταζε το Προεδρείο. Νομίζω λοιπόν ότι η σημερινή συνάντηση θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και για να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις ότι αφορά το κτίριο Μοντουάγια και το κτίριο του Στρασβούργου, αλλά και για να έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις για τους όρους ε, που αποφασίζει ίσως να εξετάσει και το ενδεχόμενο αγοράς του κτίριου Τρεμπέλ το Προεδρείο και να δούμε και ποια θα είναι η διαδικασία σε ό,τι αφορά και το συγκεκριμένο κτίριο. Θα δώσω στον εισηγητή μας πρώτα το λόγο, ο οποίος θα θέσει τα ερωτήματα και θα απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας, η Μόνικα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, σήμερα είχα πρόβλημα στον αυτοκινητόδρομο. Ε, κανονικά θα πρέπει να έχω φύγει νωρίτερα και θα μπορούσα να είχα λίγο χρόνο να μιλήσω με τους συναδέλφους, αλλά δυστυχώς ε, υπήρξε κάποιο τύχημα ε, και έχασα και το αεροπλάνο. Τέλος πάντων, ήρθα τώρα και θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη. Ξεκινάω με το κτίριο Β του Στρασβούργου. Το Στρασβούργο αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ιδιοκτήτης είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και το καλό σε αυτό το κτίριο είναι ότι το κτίριο αυτό για μας ε, βεβαίως έχει την βέλτιστη πιθανή θέση. Τα προβλήματα στο Στρασβούργο μας είναι γνωστά. Ε, στο Στρασβούργο είμαστε πολύ ε, στριμωγμένοι. Αυτό ισχύει και για τους βοηθούς, αλλά και αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον έτσι ήσυχα και ήρεμα, αν ένας ευρωβουλευτής θέλει να έχει μια ήρεμη συζήτηση με 5-6 συναδέλφους, το μόνο που του απομένει είναι το μπαρ των βουλευτών ή κάποιες άλλες ήσυχες γωνιές. Αλλά το να βρει κανείς ένα ήσυχο χώρο για ε, συζητήσεις, αυτό είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό στριμωχνόμαστε στα γραφεία μας mm. και μερικοί που μας επισκέπτονται εκπλήσονται πόσο στενά είναι τα τα μας. Το 55 ανεγέρθη αυτό το κτίριο. Από το 2007 δεν χρησιμοποιείται πλέον. Και αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ε, το είναι ο Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, που σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ λογικές ε, για μας. Μας προσφέρεται προσφέρονται 2.770 400, ε, τετραγωνικά μέτρα και θα ήμασταν ε, ευχαριστημένοι να πληρώσουμε 600 εκατομμύρια. Ενώ για άλλα κτίρια, ας πούμε για το Μονταγέ πληρώνουμε τελείως διαφορετικά ποσά. Ε, το πλεονέκτημα είναι το οικόπεδο ανήκει στην πόλη του Στρασφουργού και έχει διατεθεί για 10.000 φράγκα. Γαλλικά φράγκα. Φανταστείτε δηλαδή τίποτα, ένα τίποτα. Και αν κάποια στιγμή πρέπει να το επιστρέψουμε, θα πρέπει να επιστρέψουμε και εμείς αυτά τα 10.000 φράγκα. Βεβαίως θα υπολογιστεί διαφορετικά η τιμή του κτηρίου. Αυτό που θα είναι το πρόβλημα για μας θα είναι τα έξοδα ανακαίνιση που θα ανέλθουν σε 9,2 εκατομμύρια ευρώ. Συντήρηση, ασφάλεια, καθαρισμός και άλλα, 640.000 ευρώ το χρόνο. Επίσης το κτίριο έχει αμίαντο και η απομάκρυνση του αμοιάντου αυτό το ποσό μπαίνει μέσα στα έξοδα ανακαίνησης. Δεν έγινε διαγωνισμός, δεν προκηρύχτηκε, γιατί είναι ήδη ευρωπαϊκό ε, κτίριο και δεν υπάρχει άλλο ανταγωνιστικό κτίριο στην περιοχή. Το μόνο που θέλω να πω είναι αυτό που με ενοχλεί λιγάκι στην όλη διαδικασία είναι το εξή. Το κτίριο ίσως ήταν λιγάκι ακριβό εντάξει, αλλά η διαφορά μας είναι περίπου 100 ή 200.000 ευρώ. Αυτό είναι το επίμαχο ποσό που θα μπορούσε να υπάρξει μια έκπτωση. Σε τελική ανάλυση είναι συμπαθητικό. Εκείνο που με ενοχλεί και το ίδιο ισχύει και για το Μοντουαγέ και το λέω με κάθε ειλικρίνεια στην Επιτροπή, το κτίριο αυτό από το Σεπτέμβρη είναι έτοιμο και δεν θα έπρεπε η πρόταση να μας υποβληθεί τρεις ημέρες πριν από την ε, εκπνοή των, ε, των δυνατοτήτων που υπάρχουν, αλλά να μας έδιναν το σχέδιο της σύμβασης τον Οκτώβρη για να μπορούμε να το συζητήσουμε και να μην φτάσουμε στο παραπέντε λίγο πριν από το τέλος του έτους. Αυτό είναι δυσάρεστο. Πάω τώρα στο κτίριο Μοντουαγέ. Και εκεί έχουμε φασαρίες, πιο πολλές για να είμαι και ειλικρινής. Από πλευράς αρχής το θεωρώ απαράδεκτο το ποια ακριβώ είναι η στρατηγική των διαπραγματεύσεων. Η στρατηγική διαπραγματεύσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η απόλυτη καταστροφή. Και το λέω με κάθε ειλικρίνεια και ελπίζω η Επιτροπή να συμμερίζεται την άποψή μου. Εγώ θεωρώ ότι είναι παντελώς απαράδεικτο να έχουμε να κάνουμε με ένα και μόνο ιδιοκτήτη και να διαπραγματευόμαστε με αυτόν με τέτοιο τρόπο που να είναι και αυτό σίγουρος ότι θα παραμείνει ο ένας και μοναδικός. Όλες οι άλλες, ε, όλοι οι άλλοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν αφορούν ε, ε, μισθωτήρια συμβόλαια και παρεμφερή. Αλλά το θεωρώ απαράδεικτο ένας πολιτής ή αν θέλετε ένας εκμισθωτής που τελική ανάλυση χρεώνει και πολύ πολύ ακριβά νίκια θα έπρεπε να μας οδηγήσει στο να αναζητήσουμε εμείς και κάποιες άλλες τρεις-τέσσερις εναλλακτικέ λύσεις απλά και μόνο για να έχουμε ένα μεγαλύτερο διαπραγματευτικό ατού στα χέρια μας. Δεν το κάναμε και καταλήξαμε εδώ που είμαστε. Πρόκειται λοιπόν για ένα κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε το 1990 με συνολική έκταση 5.700 τραγωνικά μέτρα 3.700 περίπου τα τετραγωνικά ε, μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γραφεία. 250 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτή ήταν η αρχική τιμή. Και πρέπει να πω ότι η παλιά τιμή ήταν ε, υπερβολική. Καλά τους ε, ταΐσαμε τόσα χρόνια. Και βεβαιώς καλό είναι το ότι στις διαπραγματεύσεις ξεκινήσαμε από χαμηλότερη τιμή ενικίου Όμως και αυτή η χαμηλότερη τιμή είναι υψηλότερη από, τις, ε, από τα νέα μισθωτήρια συμβόλαια της περιοχής και τα νέα ενίκαια που δεν είναι 250 τετραγωνικά μέτρα, το ανώτατο είναι 240 τετραγωνικά μέτρα. Άρα δηλαδή για μας ε, αυτό, αυτή η τιμή, αυτή η προσφορά είναι υπερβολική. Η διοκτήτηση είναι η DEVA 1. Η DEVA 1 είναι μια εταιρεία ε, με χρηματοδότες από τις αραβικές χώρες. Ναι. Και ε, αυτό έχει επίσης αμίαντο. Θα υπάρξει ε, σχετική γνωμοδότηση. Δεν έλαβε χώρα ε, Δημόσιο διαγωνισμός και θέλουμε να το αγοράσουμε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τη στρατηγική πίσω από όλα αυτά. Η στρατηγική είναι όσο πιο κοντά στο Κοινοβούλιο να αποκτήσουμε κάποια κτίρια έτσι ώστε αυτοί που είναι υπάλληλοι και ε, δουλεύουν για το Κοινοβούλιο να μην αγκασμένοι να χαλάνε χρόνο και χρήμα για τη μετακίνηση, για Τραμπ και το καθεξής. Παρόλα αυτά όμως, λογικό θα ήταν το Κοινοβούλιο να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις και να μην υπάρχει μία και μοναδική λύση, γιατί αυτό το γνωρίζουν οι πολιτές. Παρότι λοιπόν ασκώ αυτή την κριτική, θέλω να συμπληρώσω ότι αν τώρα απαιτήσουμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν, λόγω των 500.000 ή το πολύ πολύ του ενός εκατομμυρίου που πληρώνουμε παραπάνω, βεβαίως γνωρίζω πολύ καλά ότι το ποσό αυτό για το φορολογούμενο ε, δεν είναι και μελιτέο, γι' αυτό και εγώ ασκώ κριτική. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι είναι σημαντικό, είναι σωστό να αγοράσουμε αυτό το κτίριο. Γιατί αν ενοικιάσουμε στην περιοχή εκεί ένα κτίριο ανεξάρτητα από το ότι στις 31 Δεκάτου εκπνέει το μισθωτήριο συμβόλαιο, αν δηλαδή αποφασίσουμε κάτι διαφορετικό, τότε θα πρέπει να οδηγήσουμε τους ε, συνεργάτες μας, ε, τους υπαλλήλους, σε αναγκαστική άδεια. Ε, εντάξει, αν θέλετε να το κάνουμε αυτό, γιατί όχι, δεν θα διαφωνήσω εγώ. Και βεβαίως ε, θέλω και να πω ότι σε αυτό το μισθωτήριο συμβόλαιο που θα υπογράψουμε θα αναλάβουμε εμείς τα έξοδα ανακαίνησης που ανέρχονται, σας είπα, στο περίπου 1,2 εκατομμύρια πρόβλεψη. Στο τέλος θα είναι σίγουρα περισσότερα. Και αυτό οδηγεί στο ότι ξεκινάμε από μια τιμή ενικιού ε, που είναι πολύ πιο πάνω από τα 260 για να μην πω 270 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με λίγα λόγια λοιπόν το, δικό, το κτίριο αυτό είναι φαρμακερά ακριβό, έχει όμως μια πολύ καλή θέση από πλευρά στρατηγικής και δεν θα αφήσω να μου το πάρουν μέσα από τα χέρια. Ε, δεν είναι καλή τιμή, αλλά αν τελικά το αφήσουμε αυτό το κτίριο, τότε θα αντιμετωπίσουμε περισσότερες δυσκολίες από το να το αγοράσουμε. Ε, έχει νόημα να το αγοράσουμε το κτίριο αυτό παρά το ένα εκατομμύριο φέση, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση και σε τελική ανάλυση για μας αυτή η λύση είναι η καλύτερη και από πλευρά στρατηγικής, ε, σας είπα, έχουμε το πλονέκτημα του ότι είναι κοντά και πολλά άλλα. Ε, και σε τελική ανάλυση με αυτή τη στρατηγική περί κτηρίων. Ε, νομίζω αυτήν ακολουθήσαμε και έτσι αγοράσαμε, νοικιάσαμε κτίρια που επιθυμούσαμε. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα δύο θέματα θα ήθελα να τα εξαντλήσουμε ε, πριν πάω στο επόμενο. Insofern wäre ich also jetzt grundsätzlich für Montoyer. Ε, σας λέω λοιπόν, είμαι κατά και ασκώ έντονη κριτική στο κτίριο Μοντουαγέ και λόγω στρατηγικής και λόγω διαπραγματεύσεων και επιμένω τουλάχιστον σε αυτή το συμβόλαιο να εντάξουμε μία ρήτρα περί επομάκρυνσης αμοιάντου. Γιατί αν τελικά εμφανιστεί και σε αυτό το ε, κτίριο αμιάντος, ε, να μην το πληρώσουμε πάλι εμείς, πρέπει να το συζητήσουμε. Και νομίζω ότι ε, ήδη αρκετά υποστήκαμε με αυτό το κτίριο λόγω της λανθασμένης στρατηγικής. Και να πω και κάτι τελευταίο. Μερικές φορές όταν είναι κανείς για ένα αυτό που τίθεται επιτάπητο είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα λαβύρινθο εγγράφων με τα οποία στόχο είναι είτε να παραπλανηθεί ο εισηγητής είτε να υπάρξουν κάποιε αλλαγέ στα χρονοδιαγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να μην μα υποβάλλετε ε, προτάσει για κτίρια που μετά από 14 μέρε εξαφανίζονται από του ηλεκτρονικού υπολογιστές. Να μας στέλνετε πραγματικά ουσιαστικές εναλλακτικέ λύσεις όπου ε, το όντι χρειάζεται χρειάζονται κάποιες επισκευές, κάποια ανακαίνιση και θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιος περισσότερος χρόνος στη διάθεση του εισηγητή. Ε, γιατί με τρόπο αυτό αποφεύγονται οι εντάσεις και εν πάση δεν είμαστε και ανόητοι για να μην μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λογική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, Madame le Ευχαριστούμε κυρία εισηγήτρια. Ο κύριος Γενικός Γραμματεύς. Κοιτάξτε, νομίζω επειδή μιλάμε για διάφορα κτίρια, αυτό που έχει νόημα είναι τα κτίρια να τα εντάξουμε στην μεσοπρόθεσμη στρατηγική μας κτηρίων. Το Προεδρείο λοιπόν αποφάσισε και η Ολομέλεια ενέκρινε ε, αντί αμφισβήτητα να υπάρχει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική κτηρίων. Αυτή εγκρίθηκε το 2010 και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής κτηρίων ε, ορίζονται λεπτομερώς και οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν λοιπόν θα αναφερθώ στις αρχές, δηλαδή αγορά, έγκαιρη αποπληρωμή του χρέους και τρίτον άμεση γυτνίαση με τα αλλακτήρια, γιατί δεν θέλουμε να βρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση ε, στην οποία βρίσκεται η Κομισιόν, η οποία ε, στη τελική ανάλυση έχει διασπείρει τα κτίρια της ολόκληρη την πόλη. Με αυτήν λοιπόν την ε, στρατηγική εντοπίσαμε συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία μεσοπρόθεσμα, και όταν μιλάμε για μεσοπρόθεσμα εννοούμε περίπου δύο χρόνια, μια στρατηγική που να, μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε δύο χρόνια χρόνια. Τώρα φτάνουμε στην κατακλίδα αυτή τη στρατηγική. Τώρα λοιπόν πρέπει να ληφθούν οι ε, αποφάσει. Αναφέρομαι στο κτίριο ΚΑΝΤ στο Λουξεμβούργο. Στι Βρυξέλλε, για τι Βρυξέλλες, αυτή τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική κτίριων ορίσαμε ότι χρειαζόμαστε επιπλέον χώρο για τα διοικητικά ε, περίπου 26.000 μέχρι 30.000 τετραγωνικά μέτρα. Και αυτό είναι το κτίριο που αναφέρθηκε, που ονοματίστηκε, είναι το κτίριο Τριμπέλ το κτίριο το οποίο είναι απαραίτητο για επιπρόσθετο προσωπικό για περίπου 10 μέχρι 12.000. Όσον αφορά το κόστος της ανακαίνησης, ε, παρότι όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τα κτίρια μας είναι καινούργια, δεν ισχύει αυτό. Το κτίριο PHS ε, δεν είναι πια καινούργιο, πρέπει να ανακαινιστεί. Επίσης και το κτίριο Eastman και η ε, ο δεύτερος νηπιακός σταθμός, πεντοβρεφονηπιακός σταθμός. Αυτά όλα θα περάσουν στην ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το θέμα του κτηρίου Μοντουαγέ 70 και έτσι εξηγείται γιατί διαπραγματευτήκαμε για το κτίριο αυτό. Διότι η στρατηγική μας πλέον είναι όχι να νοικιάζουμε κτίρια, αλλά να παραμένουμε ενοικιαστές κατ' εξαίρεση και στο μέλλον να γινόμαστε ιδιοκτήτες. Για το Στρασβούργο, στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης στρατικής κτηρίων του Μαρτίου του 2010, υπάρχει ένα κτίριο ε, το οποίο πρέπει να καλύψει και τις ανάγκες του διαμεσολαβητή. Δηλαδή ε, αυτό το κτίριο θα φιλοξενήσει τον ε, διαμεσολαβητή και έτσι θα απελευθερωθεί ένα δυναμικό τετραγωνικών μέτρων για το Κοινοβούλιο και κυρίως για τους Ευρωβουλευτές. Η στρατηγική αυτή στο πλαίσιο του προπολογισμού του 2010 χαιρετίστηκε όχι μόνο από την Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά συνολικά από το σύνολο της Ολομέλειας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που πρόκειται να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε τα προγράμματα αυτά που σημαίνει ότι εντάσσονται κάποια κτίρια σε μια στρατηγική η οποία στρατηγική δεν εγκρίνεται μόνο από το Προεδρείο αλλά από το από την Επιτροπή Προλογισμών και από την Ολομέλεια. Όσον αφορά τώρα τα τρία κτίρια μεμονωμένα. Πάμε στο Μοντουαγέ 70 καταρχήν. Το κτίριο αυτό, το Μοντουαγέ 70, είναι ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή το κτίριο αυτό το χρησιμοποιούν οι συνεργάτες μας, ε, κυρίως η Γενική Διεύθυνση Ίνλο. Και εκεί έχουν ζητηθεί πάρα πολλές γνωμοδοτήσεις ε, για την αξία του κτηρίου. Αυτά που είπε η κυρία εισηγήτρια για την πολιτική κτηρίων, δηλαδή πράγματι είμαστε στην επάνω βαθμίδα της κλίμακας των τιμών, αυτό ισχύει και κανείς δεν το αμφισβητεί. Όμως υπάρχουν κάποιοι λόγοι που οδήγησαν το Προεδρείο παρόλα αυτά να αποφασίσει υπέρ της απόκτησης αυτού του κτηρίου και οδήγησαν το Προεδρείο να λάβει και τη σχετική απόφαση. Καταρχήν λοιπόν, για μας ένα κτίριο το οποίο είναι μεσοτυχία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαφορετική αξία από ένα κτίριο το οποίο είναι 500 μέτρα ή ένα χιλιόμετρο μακριά από το κεντρικό κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παραμένουμε λοιπόν στην απόφασή μας ότι τα κτίρια είτε θα συνδέονται μεταξύ τους, είτε θα μπορούν να συνδεθούν, είτε στην ιδανική περίπτωση να χρειαστεί κανείς να διασχίσει μόνο τον δρόμο και να πάει απέναντι. Αυτό λοιπόν είναι ένα κτίριο το οποίο καλύπτει αυτό το, το κριτήριο, αυτό το το Επιπλέον, το κτίριο αυτό έχει ένα μεγάλο κήπο, ε, το οποίο ε, μπορεί να έχει μεγάλη σημασία και για άλλα προγράμματα. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό γιατί εκεί θα μπορούσε να ε, κατασκευαστεί βρεφονιπιακό σταθμός. Δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά στο λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, ε, το κτίριο αυτό έχει υπερβολικά ε, πολύ χώρο στάθμευσης και εδώ αντιμετωπίζουμε όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες. Δεν έχουμε επαρκή αριθμό θέσεων στάθμευσης. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε σε όλους τους συνεργάτες μας θέσεις στάθμευσης. Επίσης, είναι αλήθεια ότι το κτίριο αυτό ή μάλλον κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχουν πολλά κτίρια που να πολλούνται. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ λύσεις ε, στην άμεση γειτονιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εδώ συνέβη το ίδιο, δηλαδή ο ιδιοκτήτη για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν πρόθυμο να μιλήσει για πώληση, τελικά όμω ε, συνέβη κάτι τέτοιο και αυτό οδήγησε στο ότι βέβαια ο εισηγητή βρίσκεται σε ισχυρή, ο ιδιοκτήτη με βρίσκεται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Εμεί μπορέσαμε να, ή μπορούμε να αγοράσουμε το κτίριο χωρίς να ζητήσουμε επιπρόσθετα κονδύλια. Θα το αγοράσουμε από τα πλεονάσματα που θα προκύψουν στο τέλος του 2011. Το κτίριο αυτό εντάσσεται στη μεσοπρόθεσμη στρατηγική μακτηρίων δηλαδή μετάβαση από τον ενοικίαση στην ιδιοκτησία. Επίσης, πρόκειται όπως σας είπα, για ένα κτίριο που είναι μεσοτυχία με το κτίριο Αλοκασιών Φαμιλιάλ Belgian και αυτό θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να το αγοράσουμε γιατί και αυτό είναι ε, στην ίδια γειτονιά. Η βελγική κυβέρνηση αποφάσισε να ε, θέσει την Αλοκασιών Familial Στι αρμοδιότητε τη ε, περιφέρεια, τη τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι και αυτό το κτίριο θα μπορούσε να καταστεί ενδιαφέρον για μας. Η συγγήτρια ε, πρότεινε να υπάρχει μια ρήτρα για απομάκρυνση αμοιάντου ε, και αυτό θα συμβεί σίγουρα. Θα συμπεριληφθεί αυτή η ρήτρα στη σύμβαση. Για το Μπατιμόν Μπε, για αυτό το κτίριο, η συγγήτρια αποφάνθηκε λεπτομερώς. Όπως σας είπα, εκεί στόχος μας είναι να εγκατασταθεί μετά την ανακαίνιση του κτηρίου ο διαμεσολαβητής και έτσι ε, στο κεντρικό κτίριο να ελευθερωθεί χώρος, να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για τους ευρωβουλευτές. Τώρα, ποιο θα είναι το τελικό σχέδιο η χωροτέτηση. Αυτό θα αποφασιστεί, αλλά εν πάση τόσο θα ε, απλωθούμε λιγάκι στο κεντρικό κτίριο. Αυτό ισχύει κυρίως για τους ε, ευρωβουλευτές, εκείνους ε, που μοιράζονται το γραφείο τους με τους βοηθούς. Και τα λέω όλα αυτά διότι θέλω να περάσω τώρα στο επόμενο κτίριο, στο κτίριο Τρεμπέλ. Το Προεδρείο την Τετάρτη αποφάσισε το κτίριο αυτό ή το σχέδιο αυτό να υλοποιηθεί, να αγοραστεί το κτίριο Τριμπέλ. Αυτό εντάσσεται στην μεσοπρόθεσμη στρατηγική μας κτιρίων. Μιλάμε για 30.000 τετραγωνικά μέτρα και εδώ πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας ε, σε βάθος βολιτοσκόπηση της αγοράς, το αποτέλεσμα συζητήσεων και με άλλες προσφορές στο Ευρωπαϊκό ε, κοινοβούλιο. Υπάρχει μια σειρά πλέον εκτιμάτων που μπορείτε να τα δείτε και στο χάρτη. Δηλαδή, αν θέλετε, το κτίριο αυτό είναι εκείνο που κλείνει την ε, Esplanade Ζολιντανόσκ. Βρίσκεται στο κάτω μέρος, μόνο 15 μέτρα πέρα από την άλλη πλευρά του δρόμου. Είναι ένα νέο κτίριο υπό ανέγερση που σημαίνει ότι θα ολοκληρωθεί το 2017. Μιλάμε για 30.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια και ε, θα έχει την ανώτατη πιστοποίηση ε, φιλικότητας προς το περιβάλλον. 4.000 ευρώ, κάτι πάνω από 4.000 ευρώ είναι η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο, που είναι περίπου λίγο παραπάνω από την τιμή της αγοράς. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση, αντιμετωπίζουμε την εξής ιδιάουσα κατάσταση. Το βελγικό κράτος μας διέθεσε πριν από λίγο καιρό 86 εκατομμύρια, τα οποία μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν μόνο για κτίρια. Αυτά τα 86 εκατομμύρια που διαθέτουμε πρέπει να ε, διατεθούν για κτίρια. Κατόπιν τούτου, ένα μεγάλο κομμάτι πάνω από το ίμιση, δηλαδή και πάνω από τα 2 τρίτα του ποσού για την αγορά του κτηρίου Τριμπέλ θα ε, χρηματοδοτηθούν με αυτόν τον τρόπο. Και αν προσθέσουμε και άλλα 15 εκατομμύρια η προκαταβολή από τα κονδύλια ε, που θα προκύψουν από το 2011 ως πλεόνασμα. Ε, έχουμε χρηματοδότηση 101 εκατομμύρια, απομένουν μόνο 24 εκατομμύρια αυτό το ποσό ε, θα πρέπει να διατεθεί το 2017 και αργότερα. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό ποσό, το οποίο εν πάση περιπτώσει μπορούμε να καλύψουμε και με τον τρόπο αυτό θα έχει πλέον ε, αποφασιστεί οριστικά το τι ακριβώς θα κάνουμε με τα 86 εκατομμύρια που μας διέθεσε το βελγικό κράτος. Θα είναι μια πολύ λογική επένδυση αυτή που θα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά θα μπορέσουμε ε, να επιστρέψουμε στο τέλος του έτους και ένα σημαντικό ποσό στα κράτη-μέλη. Αυτό το project έχει το εξής σχέδιο. Δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι οι εργολάβοι, αλλά ένας τρίτος. Το κτίριο το αγοράζουμε με σταθερή εγγύηση, με εγγύηση σταθερών τιμών ε, και με ε, κάλυψη αστικής ευθύνης που είναι πολύ σημαντικό για μας. Νομίζω ότι σας έδωσα μια πολύ καλή εικόνα αυτών των τριών προγραμμάτων. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι ότι τα προγράμματα αυτά, ε, τα projects αυτά δεν είναι, έτσι, δεν είναι αυτοσχεδιασμός, είναι το αποτέλεσμα σχεδιασμών που κράτησαν δύο χρόνια, είναι το αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων που έλαβε όχι μόνο το Προεδρείο, αλλά και το αποτέλεσμα της υποστήριξης από την Επιτροπή Προπολογισμών και από την Ολομέλεια. Αν θέλετε τώρα ναι. βρισκόμαστε στο τελευταίο σκαλί, ε, τώρα που εκπνέει βέβαια και η θητεία αυτού του Προεδρείου, βρισκόμαστε ε, στο τέλος ε, εφαρμογής της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής. Γι' αυτό λοιπόν η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί τώρα ή στο, στο άμεσο μέλλον. Είναι, ακριβώς αυτός ο λόγος είναι και γιατί καλή καλείται η Επιτροπή Προπολογισμών να λάβει απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματεύ. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Χάγκελουντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ τη Μόνικα και πάλι για όλα όσα έχει κάνει για αυτά τα προβλήματα. Είναι και τεχνικά και οικονομικά και τελικά βέβαια πολιτικά. Επίσης ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα για την παρουσία του που θα μας βοηθήσει πολύ εδώ να λάβουμε αποφάσεις. Είναι προφανές ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα δηλαδή να έχουμε τις προτάσεις νωρίτερα από ό,τι τις είχαμε, πιο έγκαιρα. Μα εξήγησα ε, βέβαια ο γενικό Γραμματεύς του λόγου των καθυστερήσεων, αλλά παρόλα αυτά είναι θεμητή, θεμητό και το παράπονο της εισηγήτριας για τι καθυστερήσει. Είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν αυτέ οι αποφάσεις με τέτοιο τρόπο. Παρακαλώ να το λάβει υπόψη του σοβαρά ο Γενικός Γραμματεύς για το μέλλον. Γενικά νομίζω ότι πρέπει να σημειώσουμε ότι και στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη προσπαθούν οι διοικήσει να κάνουν περικοπές και οικονομίες και γι' αυτό πρέπει να δούμε αν είναι σωστό να επενδύουμε σε νέα κτίρια τα χρήματα του φορολογουμένου και της φορολογουμένης. Παρ' όλα αυτά βέβαια πρέπει να έχουμε κατάλληλα κτίρια για τη δουλειά μας. Είναι προφανές. Ίσως το κτίριο Μόντερεϊ να είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Αν και επαναλαμβάνω καθυστερημένα υπευλήθη η πρόταση. Είναι κάτι που μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Το άλλο καινούργιο κτίριο εδώ στις Βρυξέλλες είναι δύσκολο να πούμε τίποτα γι' αυτό. Ελπίζω να μην αναμένετε από εμά να πάρουμε θέση από σήμερα. Για το κτίριο του Στρασβουργού η ομάδα μου έχει συζητήσει πολλές φορές το θέμα αυτό, όπως και άλλες ομάδες σίγουρα, και έχουμε μια σαφή θέση. Δεν υποστηρίζουμε κανένα καινούριο κτίριο εν Εστρασβούργο. Γιατί θεωρούμε ότι μακροχρόνια πρέπει να σταματήσουμε να συνεδριάζουμε στο Στρασβούργο γενικώ. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε και νέα κτίρια. για την ομάδα μας τα πράγματα είναι σαφή. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ μου ο Βλαδίμηρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Γενικός Γραμματεύς θα θυμάται ότι όταν συναντηθήκαμε την πρώτη φορά ακούσαμε ανάλογα παράπονα για καθυστερήσεις υποβολής των εγγράφων και των προτάσεων. Ακόμη και όταν επρόκειτο για απλές μεταφορές χρημάτων, τα έγγραφα τα είχαμε μια-δυο μέρες πριν και είχε δεχτεί ο γραμματεύς τότε ότι είναι καθυστερημένη η υποβολή αυτή και για εκείνον. Καταλαβαίνω ότι δεν φταίει εκείνος, αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Εμείς Καμιά φορά παίρνουμε με μεγάλη καθυστέρηση μέχρι και 20 θέματα φακέλους και δεν μπορούμε εύκολα να πάρουμε αποφάσεις έτσι, υποπίεση. Εμείς πιστεύουμε ότι ως σώμα που συζητάει τον προϋπολογισμό πρέπει να έχουμε πληροφόρηση συνεχώς, μια ροή συνεχή διαρκή. Γιατί η έγκαιρη υποβολή πληροφοριών μας διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων. Όπως είπε βέβαια και κάποιος άλλος, η μόνη εναλλακτική λύση που έχουμε σήμερα είναι αυτή που μας υποβάλλεται και άμα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, τι είδους διαπραγμάτευση μπορούμε να κάνουμε. Και πώς να κρίνουμε αν η τιμή είναι λογική. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο ελιγμών λοιπόν. Αλλά τα κοινοβούλια. Ναι μεν καμιά φορά χρειάζεται επιγόντως να λάβουν αποφάσεις αλλά συνήθως σκέφτονται δεόντως τις αποφάσεις που παίρνουν πριν τις πάρουν. Γι' αυτό θα θέλαμε αφού και η Κομισιόν ζητάει όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τους κανόνες που ισχύουν για τις δημόσιες προμήθειες και εμείς το ίδιο να κάνουμε. Αν συμφωνούσαμε αν εγκρίναμε να γίνονται οι επισκευές από τους κατασκευαστές, τότε θα διαφωνούσα, θα διαφωνούσα, δεν μπορώ να το δω αυτό. Αλλά δεν θα ήθελα να θεωρήσω ότι έχουμε μπροστά μας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε. Πολλές φορές συζητούμε τα κτίρια με μία μόνο πρόταση μπροστά μας. Μία προσφορά. Ίσως θυμάστε συνάδελφοι όταν συζητήσαμε το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο το 7 ετές είχαμε πει να κόψουμε κατά 5% τις διοικητικές μας δαπάνες. Το 2005, το 2005 λέγω πριν από 7 χρόνια ακριβώς, είχε σημειωθεί τεράστια αύξηση στις δαπάνες λόγω της διεύρυνσης. 8% πιο πάνω δαπάνες για τα κτίρια για τον τίτλο 5. Και τώρα φαίνεται από τα στοιχεία ότι στο ίδιο αυτό κεφάλαιο συνεχίζουν να αυξάνονται οι δαπάνες. Άρα είναι απολύτως απαραίτητο και κατεπήγον να έχουμε περαιτέρω πληροφορίες για να ξέρουμε αν μπορούμε να αποφασίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χοχμά για την έκθεσή της και τον κύριο Βέλη για τα σχολιά της. Ό,τι αφορά το Μοντουαγέ. Αν υπάρχει αμύαντος, στο κτίριο φυσικά κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Στο Στρασβούργο νομίζω ότι το Συμβουλίο της Ευρώπης είχε θέσει το ζήτημα της φορολογίας μεταξύ 6 και 7 εκατομμυρίων Και βέβαια σίγουρα το θέμα της έδρας είναι σημαντικό. Θα παραμείνουμε μακροπρόθεσμα στο Στρασβούργο. Άρα έχει νόημα να αγοράσουμε ένα ακόμη κτίριο εκεί για το τριμπέλ από τα έξοδα μετακίνησης θα υπάρχουν κάποια κονδύλια. Ίσως λοιπόν υπάρξουν εξοικονομήσεις από το κομμάτι αυτό. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Μιλάμε για 15 εκατομμύρια έχουμε στο τραπέζι. Ίσως μπορούσαν να γίνουν κάποιες ε, οικονομίες. Thank you, Chair. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τη Μόνικα που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ήταν και ιδιαίτερα συνεργάσιμη με τις άλλες ε, πολιτικές ομάδες. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων και νομίζω ότι ήταν και ιδιαίτερα θετικά όλα όσα συζητήσαμε. Σε ό,τι αφορά του ανθρώπου μου, συμφωνώ. Ε, άκουσα τι είπε ο κύριος Μάνκα, κυρίως. Δεν θέλω να επαναλάβω, αλλά να εξηγήσω και εγώ κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε την αξιολόγηση του χώρου που χρειαζόμαστε, το πετούμενου χώρου. Χρειαζόμαστε μια τέτοια αξιολόγηση, έγινε το 2009, 40-46 τετραγωνικά μέτρα ήταν. Το 2010 είχαμε μια πιο χαμηλή εκτίμηση. Νομίζω ότι ξεκίνησε μια να αγορά στο Κοινοβούλιο και ήταν 35 με 42.000 τετραγωνικά μέτρα τότε η επιφάνεια. Ε, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που αναφέρει τώρα ο κύριος ε, Βέλη, ήταν λίγο πιο χαμηλά από αυτά. Εγώ προσωπικά, το δεν ξέρω, μπορεί να μου διέφυγε, αλλά δεν έχω δει επικαιροποίηση αυτής τη αξιολόγηση, τουλάχιστον σε έφθετο χρόνο, γιατί τι αποφάσισα που θα πρέπει να λάβουμε τώρα. Υπάρχουν γραπτό αυτά τα στοιχεία και υπήρχαν διαθέσιμα πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίε για αυτά τα κτίρια. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και αυτό δεν αφορά μόνο τι Βρυξέλλε, αλλά αφορά και το Στρασβούργο. Τι χώρο χρειαζόμαστε τελικά στο Στρασβούργο. Να σας υπενθυμίσω ότι στα ψηφίσματά μας ε, είπε παραδείγματι σε ένα ψήφισμα πολύ ξεκάθαρα τοποθετούμαστε ως εξή Η σημαντική μακροπρόθεσμη, με, μεσοπρόθεσμη στρατηγική την έχουμε, εντάξει, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, καθώς και την ανάγκη εξέτασης διαφορετικών επιλογών και εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Και νομίζω ότι έγινε και συζήτηση για την ε, περίπτωση ανοικοδόμησης κάποιων ε, εγκαταστάσεων ε, στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, ε, ξέρουμε ότι στα γραφεία υπάρχουν ντους. Αυτά θα μπορούσαν να γκρεμιστούν, για παράδειγμα, και να εξοικονομηθεί χώρος για τα γραφεία των βουλευτών. Άρα, πριν ληφθεί απόφαση για το κτίριο B, Β, έχουμε εξετάσει όλες τις παραμέτρους. Δεν είμαι πεπισμένος από αυτού. Θέλουμε περισσότερες πληροφορίες. Επίση, ένα πιο σημαντικό ζήτημα, ζήτημα αρχή, Είδα πάλι τα ψηφίσματα που έχουμε λάβει κατά καιρού στο Κοινοβούλιο, έχουμε γκρίνει το 2010, το 2011 και για το 2012 υπάρχουν τρία πράγματα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα. Πιστεύετε ότι οι προτάσεις που διατυπώνεται τώρα ανταποκρίνονται στα αιτήματα των ψηφισμάτων, σέβονται αυτά τα ψηφίσματα. Εντάξει, είπα, ζητήσαμε αυτή τη μεσοπρόθεση μακροπροστατική, την έχουμε. Αλλά υπάρχουν εναλλακτικέ δυνατότητε χρηματοδότηση. Πού είναι αυτό, δεν το βλέπουμε στο κείμενο. Και επίση, πολύ συγκεκριμένα, τα 86 εκατομμύρια που λάβουμε από την ε, βελγική κυβέρνηση. Ζητάμε πληροφορίες, λέμε, σε σχέση με αυτά τα έσοδα και εναλλακτικές ε, πληροφορίες για εναλλακτικέ επιλογές προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Αυτά τα λέμε στα ψηφίσματά μας. Έχουμε λοιπόν κάποια εναλλακτική αντί του κτίριου Τρεμπέλ. Επίσης, πάλι στα ψηφίσματα λέμε Πιστεύουμε ότι η διοίκηση θα πρέπει να αναπτύξει μια πολιτική κτήρωση σε συνεργασία με την Επιτροπή Προπολογισμών. Άρα ζητούμε να είμαστε ενήμεροι για όλες τις νέες εξελίξεις ό,τι αφορά ε, σχέδια ε, δόμησης με σημαντική επίπτωση στον προπολογισμό. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό, έτσι εκτιμώ εγώ τουλάχιστον τα πράγματα, να έρχεστε εδώ, το είπε και ο Βλαδιμίρ Μάνκα, να μας ε, δίνετε 20 διαφορετικά έγγραφα λίγες ώρες πρωτού συνεδριάσει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι σέβεστε τελικά τα ψηφίσματά μας. Θα ήθελα να ακούσω τι έχει να πει για αυτά ο κύριος ε, Βέλε. Για τον Καρ Χάγκλουντ. Το πρόβλημα το κτίριο Τρεμπέλ, ε, εξ όσων εγώ αντιλαμβάνω, ε, θέλει να αναβληθεί αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι αναπόσπαστο μια της απόφασης, της πρότασης. 15 εκατομμύρια μεταφορά πίσω. Για να μην τα χάσουμε θα πρέπει αυτό να γίνει τα Χριστούγεννα. Τέλο πάντων πριν τα τέλη του εξαμήνου. Αυτή η μεταφορά αφορά την πρώτη δόση του κτηρίου Τρεμπέλ συγκεκριμένα. Άμεση λοιπόν η σχέση μεταξύ αυτή τη μεταφορά και τη αγορά του κτηρίου Τρεμπέλ. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Αν λοιπόν δεν ληφθεί απόφαση πριν το τέλο του έτου, πάνε τα 15 εκατομμύρια, τα χάνουμε. Γι' αυτό και στην συνεδρία των συντονιστών είχα προτείνει στον πρόεδρο τουλάχιστον α έχουμε άλλη μια εβδομάδα. Δηλαδή να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα μια ξεχωριστή συνεδρίαση, να έχουμε λάβει περισσότερε προφορίε για το σχέδιο του κτηρίου Τρεμπέλ. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν απλά και έτσι να το αναβάλουμε. Χάνουμε λεφτά, χάνουμε 15 εκατομμύρια. Ευχαριστώ. Θα επανέλθω στο γνωδιάγραμμα, λέει ο πρόεδρο. Ισαμπέλ τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε θα μιλήσω με τη διπλή μου ιδιότητα, μέλος της Επιτροπής Προπολογισμών αφενός, αλλά και αντιπρόεδρος στην ομάδα εργασίας για τα κτίρια αφετέρου. Μια ομάδα εργασίας που προετοιμάζει τις αποφάσεις του Προεδρείου για τα κτίρια. Και πραγματικά χαίρομαι που είναι πάρα πολύ προσεκτική και επαγρυπνή Επιτροπή Προπολογισμών, γιατί αυτή είναι και η δουλειά της. Αλλά εφιστώ την προσοχή στο εξή μέσω πολιτικών ομάδων ή της διοίκησης του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε συνέχεια να ζητάμε επιπλέον χώρο για τους βοηθούς μας, για τους ε, ασκούμενους, για τα γραφεία μας και το καθεξής και ταυτόχρονα να αρνούμαστε ή τέλος πάντων να δυσκολευόμαστε να δημοσιοποιήσουμε την ανάγκη αγοράς νέων κτηρίων. Σίγουρα δεν είναι εύκολο αυτό το να υποστηρίξει κανείς την ανάγκη για πρόσθετες ταπάνες, αλλά πρέπει και να δούμε αν πραγματικά μπορούμε όχι να έχουμε άνεση, αλλά να έχουμε το σωστό χώρο. 18 νέοι βουλευτέ, ε, όλες οι αιτήσει και τα αιτήματα που υπάρχουν. Και ανοίγω παρένθεση για το κτίριο Τρεμπέλ. Η ιδέα είναι εκεί να τοποθετήσουμε τις διοικητικές υπηρεσίες και σε αυτό εδώ το κτίριο να μείνουν οι πολιτικές ε, δραστηριότητες, δηλαδή οι πολιτικές ομάδες, ε, οι συνεργάτες μας, έτσι θα έχουμε καλύτερο συντονισμό εργασίας. Κύριε Χολμάγερ, δίκιο έχει και ίσως και όλοι δίκιο έχουν ότι είναι ένα πάζλ. Πράγματι, έτσι έχουν τα πράγματα, δεν ελέγχουμε και ευτυχώ είναι και δική μα δουλειά. Δεν ελέγχουμε την αγορά κινήτων στι Βρυξέλλε και συγκεκριμένα σε αυτή την περιοχή. Ξέρετε, σε όλε τι μεγάλε πρωτεύουσε τα κτίρια, τα ακίνητα δεν είναι ένα θέμα το οποίο με τον σχεδιασμό το χαρταξικό λύνεται τόσο απλά. Είναι θέμα διαθεσιμότητας, στρατηγικής εργολάβων κτλ. Και θέλω να πω ότι ε, θέλω να ευχαριστήσω την Καμαδέλτα Ινγκλό η οποία προσπαθεί ακριβώς να αποφύγει ε, κάποιες ε, συνεννοήσεις μεταξύ εργολάβων. Γιατί είναι σαν να έχουν ε, βρει το κέρας της αμάλθειας εδώ με το κοινοβούλιο. Έχουμε εργαστεί εμείς πολύ στο, Προεδρείο, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα κτίρια. Θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Έχουμε λοιπόν ε, υπολογίσει λίγο πολύ ως χώρο τις 30.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι ένα λογικό νούμερο νομίζουμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούν φυσικά να γίνουν μεταξύ Επιτροπής ε, Προεπολογισμών ε, και Ιδιοκτήτη. Πρέπει να υπάρξει και ένας μεσολαβητής, ένας ενδιάμεσος. Υπάρχουν διαπραγματευτές, τους έχει δώσει εντολή το Προεδρείο και εμείς παρακολουθούμε λίγο πιο στενά τα πράγματα σε σχέση με την Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχει η τάση διαπραγμάτευση στην τιμή της αγοράς. Υπάρχουν βέβαια και μπλόφες, όπως γίνεται ναι. πάντοτε στις διαπραγματεύσεις για να περάσουν οι καλύτερε δυνατέ προτάσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κτίριο Μοντουαγιέ, πράγματι είμαστε στα όρια, ε, στην ανώτερη τιμή. Έχουμε εξηγήσει όμω ταυτόχρονα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το κτίριο, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Για το Τρεμπέλ και για το Μοντουαγιέ όμω. Πράγματι, όπω είπατε κύριε Φέρν πάρα πολύ καλά, έχουμε αυτό το θέμα με το τέλος του έτου. Σίγουρα δεν θα έπρεπε ε, να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις και καλό θα είναι να δοθεί μια παραπάνω εβδομάδα στους βουλευτές για να μελετήσουν το φάκελ. Αλλά ε, έχουμε αυτό το, το όριο το τέλος του έτους. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε να γίνει μια νέα μελέτη ε, για τις ανάγκες μας. Υπάρχει αυτή η μελέτη. Για το Στρασβούργο. Η η δική μου ομάδα είναι ίδια με τη θέση της ομάδας Άλντε. Δεν είμαστε υπέρ νέων επενδύσεων στο Στρασβούργο, γιατί η λογική μας είναι ε, η έδρα να είναι μόνο οι Βρυξέλλες. Ε, άρα θέλουμε να είμαστε συνεπείς με αυτή την αρχή. Και επειδή οι Βρυξέλλες έχουν, ή μάλλον το Βέλγιο έχει κυβέρνηση από σήμερα, έτσι, ε, και η περιφερειο... έχουμε μια περιφερειοποίηση ε, που δεν έχει ψηφιστεί βέβαια ακόμα κύριε Βέλε και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με το Βέλγιο. Ίσως παραμείνει αυτό το κτίριο ε, για, τις, ε, για τα οικογενειακά επιδόματα αλλά μάλλον πρόκειται να περιφερειοποιηθεί αυτό το, το κομμάτι των οικογενειακών επιδομάτων. Αλλά επαναλαμβάνω δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα με το Βέλγιο. Τελευταίο σχόλιο. Νομίζω ότι πρέπει εδώ στην Επιτροπή Προεπολογισμών να ζητήσουμε να δούμε και την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω ότι η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΙΝΛΟ εργάζεται ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε κοντά και με την Κομισιόν. Νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε ζητήσει να έχουμε τη στρατηγική της Κομισιόν και για τα ε, μεγάλα έργα, για την ε, αναδιάταξη στο Σούμαν και ούτω καθεξής γιατί δεν μιλάμε μόνο για τούβλα και για γραφεία, μιλάμε και για γραφεία σε κοντινή απόσταση που είναι σημαντικά για μας. Πρέπει να έχουμε ε, τη δυνατότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις με τα λόγου γνώσεως. Καλό θα ήταν λοιπόν η Κομισιόν να έρθει εδώ να μας εξηγήσει τι γίνεται πρέπει να δούμε τι γίνεται και στην Επιτροπή. Αγοράζει, πουλάει, ε, νοικιάζει, μετακομίζει. Ε, πρέπει να ξέρουμε κι εμείς για να μπορούμε κι εμείς να χαράξουμε τη δική μας στρατηγική ως Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχετε απολύτω δίκιο. Πρέπει κάποια στιγμή να ακούσουμε και την Κομισιόν, να δούμε ποια είναι η δική της στρατηγική. Σε ό,τι αφορά την ε, ανέγερση νέων ε, κτηρίων. Ο Σαλβαδόρ Γαρίγα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, μάλλον να αρχίσω από το τέλος. Αν είμαστε συνεπείς στην Επιτροπή Προπολογισμών, το πρώτο το οποίο θα πρέπει να ζητήσουμε όταν μιλάμε για επενδύσεις σε ακίνητα, είναι αν υπάρχει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Και αν εφαρμόσουμε το ίδιο για την αμυντική πολιτική, ή την ερευνητική πολιτική, γιατί να μην το εφαρμόσουμε και για την πολιτική στα ακίνητα, την πολιτική των ακινήτων. Νομίζω ότι έτσι δείχνουμε ότι είμαστε συνεπείς κάτι που ζήτησε η κυρία Ντουιρά. Δεν μπορούμε να έχουμε μια πολιτική του Κοινοβουλίου για τα ακίνητα, να έχουμε μια πολιτική ε, της Κομισιόν για τα ακίνητα και μια πολιτική του Συμβουλίου για τα ακίνητα. Εγώ πιστεύω ότι μία από τις πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να αναλυθούν από την Επιτροπή Προπολογισμών θα ήταν μια κοινή πρωτοβουλία, ο σχεδιασμός μιας κοινή πρωτοβουλίας για την πολιτική των ακινήτων για όλα τα θεσμικά όργανα. Πρέπει να κάνουμε κάποιο σχεδιασμό, ώστε τα χρήματα των φορολογουμένων να αξιοποιούν τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν και άλλα θέματα τώρα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, ε, μάλλον είναι ε, άπτονται άμεσα των αρμοδιοτήτων τη Επιτροπή Προϋπολογισμών. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα έτη οι διοικητικοί προπολογισμοί όλων των θεσμικών οργάνων θα μειωθούν. Υπάρχει ένας προγραμματισμός. Μιλάμε για πάγωμα μέχρι μείωση του προσωπικού, των προϋπολογισμών των τριών θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα λοιπόν να εξασφαλιστεί ότι το να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε κτίρια, και να υπάρχει βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά τι δαπάνε αυτών των κτίριων, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην έρχεται αυτό σε αντίθεση με την μεσοπρόθεσμη πολιτική περιορισμού των διοικητικών δαπανών των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολύ την εισηγητριά μα, γι' αυτό άλλωστε και την ορίσαμε, όπω και του προηγούμενου εισηγητέ, για να έχουμε έτσι μια συνολική εικόνα τη πολιτική ε, για τα ακίνητα. Έχω όμως ένα παράπονο ε, σε σχέση με όσους ε, συναδέλφους έλαβαν το λόγο και ο κύριος Βέλε σίγουρα θέλει να, είναι, να υπάρχει διαφάνεια, να μας δίνει όλες τις πληροφορίες. Είπε ότι μιλάμε για την τελική φάση, τελική διαδικασία δύο ετών προγραμματισμού για τα κίνητα. Λυπούμε πολύ που τόσο γρήγορα έγιναν όλα αυτά. Όπως είπε μάλιστα και κάποιος από τους ε, προηγούμενους εισηγητές, Ούτε 48 ώρες δεν έχουμε στα γραφεία μας ε, τους φακέλους. Σίγουρα έχουμε τεχνικές δυνατότητες εντυπωσιακέ και σημαντικές, αλλά πώς να διαβάσουμε αυτούς τους φακέλους τόσο γρήγορα όσο χρειάζεται. Αυτό είναι ένα παράπονο που θέλω να απευθύνω. Και το έχουμε απευθύνει πολλές φορές από την Επιτροπή Προπολισμών, ότι τελευταία στιγμή μας δίνεται τα στοιχεία. Κάτι άλλο που ισχύει επίσης είναι ότι οι πληροφορίες που μας δίνεται είναι συνεπείς με τις αρμοδιότητες Επιτροπής Προπολογισμών, συνάδει με τις αρμοδιότητες μας στον τομέα των ακινήτων. Υπάρχει πολιτική ευθύνη για την αγορά ή μια αγορά ενός ακινήτου, για την προσαρμογή στις διοικητικές ανάγκες. Αλλά αυτό τι είναι, είναι αρμοδιότητα του Προεδρείου και όχι τη Επιτροπή Προπολογισμών. Ποιο είναι ο δικό μα ρόλο, να εξασφαλίσουμε τραπετούμενη χρηματοδότηση να είναι αυτή η χρηματοδότηση σύμφωνη με τον ετησιό προπολογισμό για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Άρα να είναι αποδεκτή η χρηματοδότηση. Ο ρόλο τη Επιτροπή Προπολογισμών υπ' αυτήν την είναι απλό. Υπάρχουν πόροι. Δίνουμε του πόρου που μα ζητά το Προεδρείο. Ασκώντα πλήρη χρήση των πολιτικών του ε, ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Αλλά το Προεδρείο είναι αυτό που θα πρέπει να απαντήσει εάν αυτό είναι ανάλογα με τις ανάγκες και αν αυτό έχει μια επίπτωση στην κοινή γνώμη, αυτό δεν ευθύνει ευθύνη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Εμείς έχουμε σαρμοδιότητα την εξέβρεση πόρων και την εκπλήρωση των ε, απαιτήσεων που μας ε, ε, αποδίδει, μας αναθέτει το Προεδρείο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα, να πει μια πολιτική ομάδα αν θέλει δεν θέλει το κτίριο στο Στρασβούργο, τι να πω. αυτή που είναι στην Επιτροπή Προπολογισμών πρέπει να ξέρουν τι αρμοδιότητες έχουν. Είπα, είμαστε εδώ για να επαληθεύουμε ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για να γίνει μια επένδυση σε ένα κίνητο. Στην Επιτροπή Προπολογισμών δεν κάνουμε πολιτική για το αν θέλουμε μία έδρα ή δύο έδρες. Νομίζω ότι αυτό αντιστοιχεί ή είναι αρμοδίτητα άλλων φορέων Μήπως θα πρέπει να δούμε τελικά ποιος είναι ο ρόλος ε, των πολιτικών ομάδων. Αν μια πολιτική ομάδα ψηφίζει ε, να αγοραστεί ή να μην αγοραστεί ένα κτίριο, μήπως πρέπει να τα ξανασκεφτούμε. Εγώ δεν ξέρω τι θα έπρεπε με βάση όλα αυτά να συστήσω στη δική μου πολιτική ομάδα. Κοιτάξτε, ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο Σαλβαντόρ, ε, σίγουρα οι άλλοι συνάδελφοι ξέρουν το θέμα καλύτερα από μένα. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο για τις ε, τρεις προτάσεις για το κτίριο Μοντουαγέ. Ε, πράγματι, συμφωνώ για τους λόγους που ανέφεραν η συγγήτρια και ο Γενικός Γραμματέας, θέση και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πίστηκα τόσο πολύ ε, για το κτίριο του Στρασβούργου. Δεν ξέρω αν αυτή τη φορά θα πρέπει να δαπανίσουμε χρήματα για το Στρασβούργο, αλλά ακόμα και αν δαπανίσουμε χρήματα, δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτός ο χώρος για τους βουλευτές και τους βοηθούς. Γιατί η πρόταση είναι όχι μόνο να ανακαινήσουμε τα κτίρια των Ευρωβουλευτών, ε, καταργώντας τα ντους, παραδείγματος ε, η πρόταση λοιπόν λέει ότι θα υπάρξει αύξηση του χώρου κατά 49%. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι χρειαζόμαστε στο Στρασβούργο αυτόν τον επιπρόσθετο χώρο για, τους, ε, για, για μας. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε και άλλες ε, πληροφορίες επί του θέματος. Για το τελευταίο κτίριο θεωρώ ότι αυτά τα 15 εκατομμύρια, αν συμφωνήσουμε από αυτού, συμφωνούμε για την πρόταση στο σύνολό της. Ξέρω ότι άλλοι έχουν πει, μιλήσει για 25 εκατομμύρια, αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ ανησυχώ, ανησυχώ επίσης και για το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Γιατί φαίνεται ότι ο χώρος γραφείων που ζητείτε θα προκύψει το 2017 Όμως ε, από το 2013 ήδη χρειαζόμαστε επιπρόσθετο χώρο. Τι θα γίνει λοιπόν από το 2013 ως το 2017 ε, χρειαζόμαστε άλλη πρόταση μήπως ή μήπως θα πρέπει να βρούμε χρήματα για ένα άλλο κτίριο έστω και προσωρινά. Υπάρχουν αυτά τα εκκρεμή θέματα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω ε, να χρειαστούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας άλλη μία εβδομάδα πριν αποφασίσουμε επί του θέματος κυρίως ε, για, το, για αυτά τα θέματα. Yes, Chairman, just brief. Ο Κάρχαν μου ζήτησε συγγένει συντομία το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, να πω απλά ότι από το πρίσμα όσων ακούστηκαν και εμείς στηρίζουμε την ανάγκη να συνεδριάσουμε εκ νέου για να επανεκτιμήσουμε το θέμα του κτηρίου Τρεμπέλη. Χέλγα Τρούπελ. Έχοντας ακούσει τους ε, συναδέλφους, ε, θέλω να κάνω μια δήλωση και να υποβάλω και μια ερώτηση. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Σαλβαντόρ ε, σχετικά με τη θέση της Επιτροπής Προϋπολογισμού γιατί ακόμα και αν είμαστε οι αρμόδιοι, εμείς δεν διαχειριζόμαστε μόνο ε, αριθμούς, τίθεται πάντα και το πολιτικό ζήτημα. Ως λοιπόν ευρωβουλευτές ε, φέρουμε και σε αυτό το θέμα την ευθύνη. Βεβαίως και είναι απόλυτα σαφές ε, ότι περνάει, εκπέμπουμε ένα πολιτικό μήνυμα όταν φασίζουμε το τι κάνουμε με τα κτηριά μας και με όλα αυτά για τα οποία είμαστε αρμόδιοι. Όσον αφορά λοιπόν το Στρασβούργο, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη δική σας την άποψη κύριε Πρόεδρε, με αυτά που είπατε στην προηγούμενη συνάντηση, ότι θα ήταν σκόπιμο να δώσουμε τη δυνατότητα στη γαλλική κυβέρνηση να υποβάλει μια άλλη πρόταση, δηλαδή να μην τους ε, στριμώξουμε σε μια κατάσταση, να μην τους ε, στριμώξουμε στον τοίχο αν υπάρχει κάποια ελπίδα να μετακινηθούν, θα ήταν λάθος να τους πρόξουμε σε λάθος ε, κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε κάποια άλλη λύση. Και αυτά τα λέω, αν υπάρχουν ε, βέβαια κάποιες ελπίδες, έστω αμυντρές, ότι μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση της η γαλλική κυβέρνηση. Και έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Βέλε, ο Σαλβαντόρ είπε ότι κατά τους επόμενους μήνες, ακόμα και αν δεν μας αρέσει, είναι πολύ πιθανό να ε, παγώσει ή να περιστεί ο προεπλογισμός ε, για θέματα διοίκηση. Και είπατε ότι το τριμπέλ θα είναι έτοιμο το 2017. Δείτε λοιπόν το εξή ερώτημα ποιες είναι οι υπόλοιπες δαπάνες που θα προκύψουν ας πούμε από τη συντήρηση του κτηρίου. Αυτές τις δαπάνες τις έχετε υπολογίσει και αν δεν τις έχετε υπολογίσει μαζί με την μεσοπρόθεσμη στρατηγική κτηρίων θέλουμε να γνωρίζουμε τι θα συνεπάγονται όλα αυτά για τον προπολογισμό μας. Μήπως ε, τεθούν σε κίνδυνο άλλα στοιχεία του προπολογισμού. Ο Γενικό Γραμματέα έχει το λόγο. Πολλά ήταν τα σχόλια, πολλέ ερωτήσει. Κλάου, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, λοιπόν, ε, ο κύριο Χακλούντ κατέστησε σαφές ότι η δική του η πολιτική αμάδα είναι κατά ε, των επιπρόσθετων κτίριων στο Στρασβούργο για λόγους αρχής. Αυτό όμως είναι μια πολιτική θέση και δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Το Προεδρείο αλλά και η διοίκηση συνεχίζει να εργάζεται με βάση την κατάσταση που υπάρχει τώρα και με βάση τις ε, διοικητικές μας ανάγκες. Εγώ δεν άκουσα κριτική ως προς το κτίριο ή ως ε, προς τις ε, προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν το κτίριο αυτό ήταν καθαρά πολιτική θέση που βεβαίως κάθε πολιτική ομάδα έχει τη δική της θέση. Ο κύριος Μάνκα είπε για άλλη μια φορά ότι πρέπει να τηρήσουμε τις διαδικασίες και αυτό το πράττουμε. Και για αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε χρόνο. Η βολιντοσκόπηση, η έρευνα αγοράς που κάναμε χρειάζεται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ε, και αυτό απαιτείται και για την στρατική κτηρίων. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικέ λύσεις. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση ενός κτηρίου που ήδη χρησιμοποιούμε, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να έρθουμε σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη και να ε, καταλήξουμε σε μια διευθέτηση. Ο κύριος ε, Χακλούντ επισήμανε επίση ότι ε, προφανώς με τη μεταφορά θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε χρήματα τα οποία αλλιώς θα προβλέπονταν για ταξίδια. Η αλήθεια είναι όλοι μας έχουμε διαπιστώσει ότι οι δαπάνες ταξιδίων των ευρωβουλευτών είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που είχαμε υποθέσει γιατί πολλοί ευρωβουλευτές ε, δεν ταξιδεύουν business αλλά με εισιτήριο που ταξιδεύουν economy και είναι ευχαριστημένοι. Έτσι λοιπόν, αν ε, προέκυπτε ή αυτό που πολλοί φοβόντουσαν ότι με το νέο καθεστώς ε, θα υπήρχε έκρηξη δαπανών, ε, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ο κύριος Φέρν έθεσε μια σειρά ερωτημάτων, καταρχήν όσον αφορά τις ανάγκες. Οι ανάγκες λοιπόν διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της ε, μεσοπρόθεσμης στρατηγικής κτηρίων το Μάρτιο του 2010. Αυτό το μέγεθος ε, είναι για μας ε, το σημείο κίνησης. Βεβαίως έχει και ο κύριος Ευρωβουλευτής που λέει όμως τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν, μπορούν να μετακινηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Στη δική μας την περίπτωση πρέπει να πούμε ότι οι ανάγκες αυξήθηκαν με τον επιπρόσθετο συμπληρωματικό προπολογισμό του 2011, τον προπολογισμό του 2000, το συμπληρωματικό του 10, τον κανονικό του 11 και την Κροατία. Αν υπολογίσετε το προσωπικό που υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό ε, στο, στην απόφαση του Προεδρού. Μιλάμε δηλαδή για άλλους 500 ε, συνεργάτες που θα προσθετούν. Αυτό αφορά τις πολιτικές ομάδες, τη διοίκηση, αφορά την Κροατία και εκεί δεν έχει υπολογιστεί και το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των βοηθών. Άρα δηλαδή ο υπολογισμός των αναγκών ε, που έγινε το Μάρτιο του 2010 κινείται περισσότερο προς τα κάτω και όχι ανωδικά. Στην ε, καθημερινή σας ε, ζωή και πραγματικότητα μπορείτε εντωμεταξύ να δείτε πόσο φορτωμένα είναι τα κτίρια μας. Την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε το απόλυτο ρεκόρ. 16.000 άτομα βρίσκονται σε αυτό το κτίριο. Είμαστε δηλαδή σαφώς πάνω από το μέγιστο δυναμικό αυτών των κτιριών. Και αυτό το βλέπει κανείς στους διαδρόμους, στις καντίνες, στα σανσέρ. Βλέπει κανείς ότι είναι μία κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί όπου είτε θα περιορίσουμε ρίζικα τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται στα κτίρια ή εναλλακτικά θα πούμε ότι θα προσφέρουμε επιπρόσθετες δυνατότητες. Πραγματικά είμαστε τελείως εκτός του αποδεκτού, εκτός του λογικού εκτός αυτού που επιτρέπει να δουλεύει κανείς αυτό το κτίριο αποτελεσματικά. Εσείς θέσατε ε, το ερώτημα κατά πόσον ε, το Προεδρείο εξέτασε εναλλακτικέ λύσεις στο κτίριο Τριμπέλ. Το πράξαμε αυτό. Είχαμε μια σειρά προσφορών ε, που εξετάστηκαν και περιορίστηκαν. Στο τέλος είχαμε τρία και μετά πάλι δύο και το αποτέλεσμα ήταν αυτό το κτίριο Τριμπέλ λόγω της θέσης του, όπως σας είπα, γιατί είναι νεόδμητο, γιατί ε, θα προσφέρει τις καλύτερες ε, προδιαγραφές ε, περιβάλλοντος και θα είναι άμεσα συνδεόμενο με τα κεντρικά κτίρια του Κοινοβουλίου. Προς ενημέρωσή σας, το Προεδρείο προσπαθεί, προσπαθεί στο βαθμό του δυνατού να σας ενημερώνει έγκαιρα. Η συγγήτρια για τα κτίρια είναι μόνιμα προσκεκλημένοι στην ομάδα εργασίας για τα κτίρια όπου προσφέρονται οι τελευταίες πληροφορίες, οι πιο επίκαιρες. Βεβαίως τα πράγματα αλλάζουν και βραχυπρόθεσμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι πρόθυμος ε, να έρχομαι πιο συχνά σε εσά, αν το θέλετε, να σας ενημερώνω για το ποια είναι η κατάσταση. Και με τον τρόπο αυτό θα είναι καλύτερα ενημερωμένη η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Όσον αφορά τώρα ε, το χρόνο που μας προσφέρεται, επουδενή δεν πρέπει να ζητάμε να ληφθεί η απόφαση μέσα σε δύο ημέρες. Ε, είναι σαφής ο κανονισμός του προϋπολογισμού και ο δημοσιονομικός, δηλαδή ο κανονισμός λέει με βάση το άρθρο 197 ε, μπορεί η Επιτροπή Προπολογισμών να αποφασίσει μέσα σε δύο εβδομάδες και όσον αφορά τα θέματα ε, Μοντουαγέ και Μπατιμόμπε, στις 21 Νοεμβρίου πήρατε τα απαραίτητα στοιχεία. Εκεί είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο. Όσον αφορά το κτίριο Τριμπέλ, τα στοιχεία σας εστάλησαν πράγματι την περασμένη Πέμπτη. Ε, είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθεί σήμερα η απόφαση σε αυτή τη συνεδρίαση και γι' αυτό ε, θεωρώ ότι και τα μέλη της Επιτροπής αλλά και εγώ θα ε, καλοβλέπαμε μια ειδική συνεδρίαση έξτρα στο Στρασβούργο για να δούμε με την ησυχία μας όλα αυτά τα θέματα και ενδεχομένως εκεί να καταλήξουμε σε απόφαση. Κυρία, η κυρία Ντιρόν ε, μίλησε ως μέλος του Προεδρείου και ως μέλος της Επιτροπής Προπολογισμών. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα σε αυτά που είπε. Ο κύριος Καρίγκα μίλησε για το κόστος. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε κατά νου ότι η αγορά κτηρίων οδηγεί σε εξοικονόμηση δαπανών. Και θα ήθελα να φέρω δύο στοιχεία από τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Κτηρίων του Μαρτίου του 2010. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι εάν υπάρξει πρόορη αποπληρωμή του ποσού, και το κάναμε αυτό, εξοικονομήσαμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 360 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω είναι σημαντικό το ποσό. Άρα δηλαδή πρόορη αποπληρωμή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ελάφρυνση του προπολογισμού και του φορολογούμενου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, στα κτίρια όπου είμαστε ιδιοκτήτες, αν αυτά έπρεπε να ενοικιαστούν και αυτό είναι ένα στοιχείο από την στρατηγική κτηρίων του 2010, θα καταβάλαμε 162 εκατομμύρια ευρώ ετησίως με τη μορφή μισθώματος. Δηλαδή αυτό θα ήταν η σημαντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού μας. Ως εκ τούτου η πολιτική, ε, την οποία θεωρεί πολύ σημαντική η Επιτροπή Προϋπολογισμών, δηλαδή να είμαστε ιδιοκτήτες, να μεριμνούμε για ουσιαστική ελάφρυνση του φορολογούμενου αλλά και του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούμε και γι' αυτό το λόγο το Προεδρείο επιθυμεί να συνεχίσει να εφαρμόζει αυτή την πολιτική. Και αν θέλετε, αυτή είναι μια απάντηση ε, προς την κυρία Τρούπελ που είπε ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία. Μα κάνουμε οικονομία. Ε, το περασμένο φθινόπωρο ε, για πρώτη φορά στην ιστορία του Κοινοβουλίου μειώθηκαν οι δαπάνε κατά 25 εκατομμύρια παρότι είχε εγκριθεί το σύνολο των δαπανών από το Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να κάνουμε οικονομία ε, κατόπιν του, αυτά που σας προτείναμε δεν είναι αντίφαση με την πολιτική μας και εξάλλου αυτή την πολιτική όχι μόνο τη στηρίζουμε αλλά η πολιτική αυτή προβλέπεται, απαιτείται κιόλα από εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τώρα, ε, έξοδα δαπάνης συντήρησης για το κτίριο Τριμπέλ. Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση της κυρίας Τρούπελ 56 ευρώ το τετραγωνικό για συντήρηση και αποκατάσταση. Πολύ χαμηλό κόστος ε, ενέργειας ε, λόγω των προδιαγραφών που ανέρχεται σε 20 ευρώ ανά τετραγωνικό. Très Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενικέ Γραμματεύ και συγγνώμη που σας κρατήσαμε παραπάνω από όσο προβλεπόταν. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα μας λείπει ο χρόνος γιατί έχουμε και άλλο σημαντικό θέμα και επί τις ψηφοφορίες. Για να ακούσουμε λοιπόν τον εισηγητή. Προτείνω το εξής. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μεν έτοιμοι να ψηφίσουμε σήμερα για το Μοντουαγέ, αλλά χρειαζόμαστε δύο ακόμη αποσαφηνήσεις στη θέση των σοσιαλιστών για το Στρασβούργο και τι θα γίνει με το Τρεμπέλ. Μετά από τη συνάντηση των συντονιστών στις αρχές του απογεύματος, ρώτησα αν μπορούμε ε, την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο να βρούμε μια αίθουσα για να το συζητήσουμε και μου είπανε ναι. Προτείνω λοιπόν να αναβάλουμε το τέλος της συζήτησης και την ψηφοφορία για τα τρία κτίρια στο Στρασβούργο για να μπορέσουμε να έχουμε εκεί μια συνολική άποψη και μια λογική ψηφοφορία. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα για τις αποσαφηνήσεις του. Χρειαζόμαστε κι άλλες πληροφορίες, ιδιαίτερα για το Τρεμπέλ. Για το Τρέμπελ επίσης ξέρουμε ότι πρέπει να ληφθούν δύο αποφάσεις σε διαφορετικές στιγμές, δηλαδή τη μεταφορά και εδώ όπως υπόθηκε το θέμα είναι αν θέλουμε να κρατήσουμε 15 εκατομμύρια περισσεύματα ή όχι, αν δεν τα κρατήσουμε τότε θα επιστραφούν στα κράτη-μέλη. Δεν θα αποφεληθεί το κοινοβούλιο δηλαδή. Αν τα κρατήσουμε τότε σε δεύτερη φάση τον Ιανουάριο ίσως μπορούμε να αποφασίσουμε. Προτείνω όμως και για τα τρία κτίρια να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Συμφωνείτε κυρία εισηγήτρια. Συμφωνώ απόλυτα. Τότε πράγματι ε, μπορούμε να συζητήσουμε και για τα τρία θέματα και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω και εγώ τα εξή. Καταρχήν, ευχαριστώ θερμά τους συνεισηγητές μου, οι οποίοι με ενθάρρυναν ε, να λέω τη γνώμη μου, οποτεδήποτε αισθάνθηκα κάποια μηχανία. Κύριε Γενική Γραμματέα, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι θέλετε να στηρίξετε τη διοίκηση. Όμως, ε, αν δει κανεί τον αριθμό των εγγράφων και χαρτιών που πήρα για το θέμα των ε, κτηρίων και τα οποία μάλιστα πολλές φορές μέσα σε δύο ημέρες τροποποιούνται ε, σίγουρα τροποποιούνται στο χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων. Αυτά θυμούνται οι συνάδελφοι Χάκλουν και ε, άλλοι που τους πίεζε ότι ξέρετε πρέπει να αποφασίσουμε για το κτίριο Μοντογέ και πάρα πολλά άλλα. Εμάς δεν μας ενημερώσετε καν ότι αποσύρθηκε ένα project που υπήρχε κατόπιν τούτου ε, θα έπρεπε έτσι να δείχνετε κάποια κατανόηση ε, για την εισηγητρία και τους ε, συνεισηγητές. Γιατί πραγματικά ήμασταν πολύ καλοπροαίρετοι απέναντι σε όλη αυτή την, θα μου επιτρέψει να το πω, χαοτική οργάνωση αυτού του θέματος αυτό που, ο τρόπος που τις συνεργασίες πραγματικά μας έφτασε λίγα στα όρια της ε, υπομονής μας και της αποτελεσματικότητάς μας. Όσον αφορά τώρα το κτίριο Τριμπέλ, πράγματι θα πρέπει να υποβληθούν κάποιες ε, ερωτήσεις, διότι αν αγοράσουμε το κτίριο, ο πολιτής ε, έχει ε, μίσθωση leasing 99 ετών. Άρα δηλαδή τι σημαίνει εδώ αγορά. Ποιες θα είναι οι οικονομικές ή οι νομικές επιπτώσεις. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα ε, που αφορούν την ουσία της ε, σύμβασης ε, και θα ήθελα αυτά λιγάκι να διευκρινιστούν. Ελπίζω, Πρόεδρε, όλα αυτά να γίνουν μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να παρακαλέσω τους ε, συναδέλφους. συνάδελφος Τρούπελ πολύ σωστά έθεσε το ερώτημα της συντήρησης. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο μιας γνωμοδότησης ε, πρωτοβουλίας να διευκρινίσουμε ε, κάποιες ε, θέσεις. Εγώ αυτό θα το παρουσιάσω ως παράρτημα, ως δική μου γνωμοδότηση στο, ε, στην Ολομέλεια. Ως Κοινοβούλιο πράγματι πρέπει να ε, σκεφτούμε τι θα γίνει με την συντήρηση. Εντάξει, δεν θα έχουμε νίκη, όμως θα έχουμε έξοδα συντήρησης και ανακαίνησης. Η Κομισιόν ε, προτείνει άλλη στατική, προτείνει μισθωτήρια συμβόλαια. Βέβαια τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι πολύ δαπανηρά και τώρα στις Βρυξέλλες ε, δεν έχει ξεκαθαριστεί τι προτείνεται να κάνει η Κομισιόν. Υπάρχει κατόπιν και η Επιτροπή των Περιφερειών που και αυτή έχει ανάγκες κτηρίων. Γι' αυτό λοιπόν σε μία έκθεση πρωτοβουλίας πρέπει ακριβώς να αναφέρεται τι προτείνει η Επιτροπή Προπολογισμών έχοντας κατά νου τα οικονομικά. Ο συνάδελφος Γκαρίγκα είπε ότι ε, θα πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε και κάτω από το πρίσμα της ε, λογικής ε, και της ε, διοίκησης. Σε τελική ανάλυση λέει όλοι οι θεσμοί θα πρέπει να έχουν μια στάση και όχι ο καθένας να ακολουθεί το δικό του τον δρόμο. Εγώ λοιπόν θα τρέψω πολύ λογικό την επόμενη εβδομάδα να λάβουμε την απόφαση. Όσον αφορά την μεσοπρόθεσμη πολιτική κτηρίων, απευθύνομαι προς τον κύριο Φέρν, πρέπει να σας πω ότι την Πέμπτη δεν μας τα στείλαν τα έγγραφα. Εμείς πήγαμε και τα πήραμε. Μας τα έστειλαν ε, επίσημα την Παρασκευή. Και ένα τμήμα των ε, εγγράφων που τα πήραμε την Πέμπτη, εκεί ε, πρέπει να σας πω ότι αναγκαστήκαμε μέχρι το βράδυ να δουλέψουμε για να σας στείλουμε και εμείς ηλεκτρονικά τουλάχιστον για άλλα κτηρία υπήρχε κάποια ηλεκτρονική ενημέρωση και γι' αυτά στο παράρτημα 2 υπάρχει έτσι μια γενική εικόνα για τις ε, ανάγκες ε, χώρου. Θα ήθελα λοιπόν επίση να πω ότι ο συνάδελφο κύριο Μάνκα πήρε αυτά τα στοιχεία, ούτε και εγώ μπόρεσα να τα αναλύσω, γιατί σα λέω ότι ήταν όλα πάρα πολύ βραχυπρόθεσμα. Ε, προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, όμω ε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Ο Γενικός Γραμματέας πολύ σωστά μας είπε τι συνεπάγεται για μας με τη μορφή πλεονεκτήματος σε η πρόορη εξόφληση χρέους. Κοιτάξτε, ε, σήμερα έχουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τα 1,3 εκατομμύρια τόκοι που θα προέκυπταν για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της τήρησης απλώς της κανονικής προθεσμίας αν όμως πληρώσουμε νωρίτερα έγκυρη και πρόωρη εξόφληση, τότε όπως σας είπα θα εξοικονομήσουμε 1,3 εκατομμύρια και γι' αυτό σας παρακαλώ να συμφωνήσετε σε αυτήν την απόφαση. Ε, και θα ήθελα ε, να ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα που έχει το θάρρος να έρθει εδώ για να ακούσει τα παράπονά μας σχετικά με την έλλειψη χρόνου. Ευχαριστώ και ε, αποχαιρετώ τον Γενικό Γραμματέα. Να πω ότι για αυτό το θέμα. Θα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση την προσεχή Δευτέρα στο Στρασβούργο στην αίθουσα SDM. Τέλο πάνω στο κτίριο SDM, στην αίθουσα 5. Θα σας ε, σταλεί και mail από τις 9 έως τις 10.30 το βράδυ, με 11 γλώσσες. Μόνο και μόνο για αυτό το θέμα θα είναι η έκτακτη αυτή συνεδρία και έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε την τελική μας απόφαση για την πολιτική των ακινήτων για το πρώτο ίμιση τη κοινοβουλευτική περίοδου, του Πρόεδρου Μπούζεκ δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους και την εισηγητρία και σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 7. Σημείο 7 της ημερησίας διάταξης. du bâtiment à la fusion nucléaire. Mes chers collègues, vous... Αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER. Un peu de calme, s'il vous plaît. Euh, nous avons... Έχουμε επιμείνει πολύ στι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό του 2012 να μην είναι περίπλοκες αυτές οι διαπραγματεύσει. Ούτε να μολυνθούν, αν θέλετε, από τη συζήτηση για την χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά την υπέρβαση κόστου για το πολύ σημαντικό αυτό ερευνητικό πρόγραμμα ITER. Και καταφέραμε να είναι ξεχωριστές οι διαπραγματεύσεις. Από την πρώτη μέρα είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε παράλληλες διαπραγματεύσεις, δύο τρένα δηλαδή που κινούνται σε παράλληλες τροχές, αυτή είναι η εικόνα έτσι που ε, χρησιμοποίει αυτή η παρομοίαση. Ε, φτάνει το 12 ε, το πρώτο τρένο στο σταθμό και μετά βλέπουμε αν μπορεί να φτάσει στον προορισμό του και το τρένο Ίτερ. Δύο τριμερείς διάλογοι έγιναν διαδοχικοί για το ίτερ. Ο δεύτερος επέτρεψε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο επίπεδο των αντιπροσωπιών. Το Συμβούλιο το εκπροσωπούσε η Πολωνική Προεδρία και την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Όπως βέβαια συμβαίνει σε κάθε τριμερή διάλογο, είναι ένας, ε, μια συμφωνία αντρεφερέντουμ. Ο Ράιμερ Μπέγκε θα μας παρουσιάσει τις, ε, τους όρους της συμφωνίας. Θα ψηφίσουμε και στη συνέχεια και θα δούμε αν υπάρχει πλειοψηφία. Οπότε θα μπορούσαμε στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε την προσεχή Τρίτη, 13 του μήνα, και έτσι να γίνει και η σχετική ε, ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Ο Ράιμερ έχει το λόγο. Ähm, Θα ήθελα να προσθέσω ότι την Πέμπτη το πρωί, την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Τριμερούς, έλαβε χώρα και συνεδρίαση των συντονιστών, όπου μιλήσαμε για τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης. Εκ των υστέρων λοιπόν αποδείχτηκε απόλυτα σωστό να διαχωριστεί να διαχωριστούν διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό του 2012 από την αναθεώρηση ε, του προγράμματος ITER. Σε τελική ανάλυση αυτό που ενδιαφέρει είναι η εκτονιστέρων των χρηματοδότηση του ITER να γίνει σε τρεις φάσεις. Στην Τριμερή Επιτροπή ο πρόεδρος και εγώ ε, συμμετείχαμε και ο κύριος Χάκλουν και ο Καλφίν ε, και στο τέλος όλοι οι μετέχοντες συμφώνησαν με την κοινή δήλωση. Ε, βλέπετε λοιπόν στο σχέδιο της έκθεσης, στο παράρτημα, την κοινή μας δήλωση στην οποία προβήκαμε την 1η Δεκεμβρίου. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι ε, σε, το, σε αυτή τη δεύτερη στάνση της ε, Τριμερός ε, το Κοινοβούλιο εμφανίστηκε με τις τροποποιημένες του προτάσεις που αφορούσαν τον προηγούμενο ε, τρίλογο, στην προηγούμενη τριμερή, η οποία διεκόπη. Μιλάμε για 1,3 δις ε, εκ των υστέρων ανάγκη χρηματοδότησης, 100 εκατομμύρια ήδη στον προπολισμό του 2012. Άρα δηλαδή αυτό που αναφέρεται στα Combi News, ε, τα 310 είναι λάθος. Είναι τα 300 εκατομμύρια από το 2012. Το δεύτερο είναι το εξής. Πράγματι, εμείς ήμασταν πρόθυμοι. Το ανώτατο όριο του κατηγορίας Α1 για τα έτη 2012 και 2003 να τα αυξήσουμε κατά 340 εκατομμύρια επιμεριζόμενα σε 650 το 12 και 190 το 13 και όπως ε, συμβαίνει στην αναθεώρηση να υπάρξει αντιστάθμιση ε, στις υποχρεώσεις ε, στον τομέα 2 και στον τομέα 5 340 εκατομμύρια για το 2011 και 174 εκατομμύρια για το 2012. Αυτό λοιπόν το μείγμα προέκυψε απλά και μόνο διότι το Συμβούλιο υπήρξαν κάποιες αντιπροσωπείες που εξακολουθούν να έχουν σημαντικά προβλήματα στο να αυξηθούν τα ποσά στον τομέα 2 για ευνόητους λόγους. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στον προπολογισμό του 2011 το περιθώριο του τομέα 2, το περιθώριο είναι κατά πολύ, μεγαλύτερο από αυτά τα ποσά. Για μας ήταν σημαντικό σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής να πούμε ότι την ημέρα κατά την οποία ψηφίζουμε για τον προπολογισμό του 2012 δεν μπορούμε την ίδια μέρα να άρουμε την απόφασή μας. Ε, δηλαδή να ενταχθεί, μάλλον το θέμα του αποθέματος δεν έπρεπε να τεθεί εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα και ε, συμφώνησαν όλοι. Κατόπιν, όσον αφορά την τρίτη φάση, δηλαδή τα 360 εκατομμύρια, τα οποία χρήζουν διευκρίνηση στις υποχρεώσεις πληρωμών. Εκεί συμφωνήσαμε οι πιστώσεις αυτές στο πλαίσιο του προπολογισμού του 2003 να εξευρεθούν και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μας είναι στο κείμενο να αναφέρεται ότι θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη και θα χρησιμοποιούνται οι διατάξεις της 17ης Μαδίου του 2006. Και ο συμβασμός λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω περαιτέρω αναθεώρηση του προγράμματος ΙΤΕΡ σε σχέση με το πολιτέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, η Κομισιόν πρότεινε 300 εκατομμύρια redeployment στο 1α, ε, τουλάχιστον 100 για τα joint undertakings. Εμείς είπαμε ότι αυτό δεν το δεχόμαστε, δεν συμφωνούμε. Και γίνεται καθαρή αναφορά στην κατηγορία 1α, αλλά αυτό δεν εμφανίζεται στο κείμενο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι οι κόκκινες γραμμές που είχαμε ορίσει, αυτά που μας είχαν πει δηλαδή οι εμείς τα τηρήσαμε και τα περάσαμε κατά κάποιον τρόπο. Και εάν τώρα κάποιες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο ε, είχαν πρόβλημα με το να αναφέρεται ο δημοσιονομικός κανονισμός γιατί υποτίθεται ότι με τον τρόπο αυτό ανοίγουν ε, κάποια παράθυρα ε, πρέπει να πω ότι ήταν, υπήρξαν αντιπροσωπείες οι οποίες αναφέρθηκαν στο ότι στο νομικό κείμενο γίνεται αναφορά στα άρθρα 21 μέχρι 23 της Διαθεσμικής Συμφωνίας. Τα όλα είναι πραγματικά ε, περίεργη συμπεριφορά και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εμείς δεν κατορθώσαμε να επιτύχουμε προσαρμογή ε, της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνθήκη της Λισαβόνας γιατί υπήρξε σύγκρουση με το Συμβούλιο και έτσι και αλλιώ ε, παραμένουν τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, δηλαδή η συνέχεια της νομολογίας εξαιρουμένων των άρθρων, τα οποία καταπίπτουν λόγω της θέσης ισχύ της συνθήκης. Η μονόπλευρη δέσμευση του Συμβουλίου στο θέμα κατά πόσον στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 003 θα πρέπει στο μέλλον να υπάρχει ομόφωνη συμφωνία ή κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πλειοψηφία, ξέρουμε ότι από αυτού υπάρχουν διαφορετικές νομικές ερμηνείες των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η μονομερής δέσμευση ε, την οποία ε, απαιτεί το Συμβούλιο. Επ' αυτού γνωρίζετε τι συμβαίνει, αλλά το να αρνείτε να γίνεται αναφορά στο κείμενο σε αυτές τις παραγράφους που είναι απλά αναπόσπαστο τμήμα των ε, συμβάσεων και ισχύουν, αυτό αγγίζει τα όρια της γελιότητας. Λυπάμαι που το λέω και κατά τα άλλα Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και παρηγοριέμαι με αυτά που είπε ο Άντερναουρ κάποια στιγμή ότι ζούμε όλοι κάτω από τον ίδιο ουρανό αλλά δυστυχώς δεν έχουμε όλοι τον ίδιο ορίζοντα. Αυτή είναι η παρηγοριά μου. Κατά τα άλλα, κύριε Πρόεδρε, αν θέλουμε να δώσουμε κάποια ευκαιρία στο πρόγραμμα ITER, και έχω την εντύπωση ότι αυτό το επιθυμεί η πλειοψηφία ε, του Κοινοβουλίου. Θα παρουσιάσουμε ένα αποτέλεσμα σε τρεις φάσεις. Αυτή ήταν η μόνη δυνατότητα να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση και κατά κάποιον τρόπο μπορέσαμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου μέσα από την Επιτροπή Προπολογισμών. Ε, το αποτέλεσμα λοιπόν των διαπραγματεύσεων είναι ικανοποιητικό, είναι ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καλούν βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τα 360 εκατομμύρια στο πλαίσιο του προπολογισμού του 2013. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι για να μην υπάρχουν διστάμενες απόψεις για το πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε για, τα, για τις ε, κοινοπραξίες, τα joint undertakings ε, και οτιδήποτε άλλο, Θέλω να σας πω ότι 460 εκατομμύρια συνδέονται άμεσα με πλήρη διαφύλαξη ε, της δημοσιονομικής ε, πειθαρχίας ε, και της, της στήρησης των συνθήκων. Δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε το δικαίωμα γνωμοδότης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα ήταν σκόπιμο Αυτά ε, να τα συζητήσουμε. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής μας και ο επικεφαλής ε, της Επιτροπής ε, Διαπραγματεύσεων προτείνει την έγκριση δύο τροπολογιών που καθιστούν αυτή τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις απέναντι στο Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της τριμερούς θέλουμε να πούμε ότι πράγματι υπήρξε πνεύμα συνεργασίας και αυτό πρέπει να το προβάλλουμε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κουκόψκι, ε, πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών, την Πολωνική Προεδρία, αλλά και τον Υπουργό Ντομινίκ, ε, για την ε, πολύ ρεαλιστική στάση τους ε, και τον τρόπο που καθοδήγησαν τις διαπραγματεύσεις που δεν ήταν εύκολο λόγω της στάσης του Κοινοβουλίου και λόγω των δικών της κανοντήτων μπορέσαμε σήμερα να σας υποβάλουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχετε μπροστά σας. Ευχαριστώ. Τα αποτελέσματα αυτά νομίζω ότι είναι τα καλύτερα ή τα λιγότερο άσχημα που θα μπορούσαμε να πετύχουμε σε αυτό το δύσκολο θέμα. Θα θυμάστε ότι πέρυσι κοντέψαμε να έχουμε συμφωνία. Τελικά δεν επετεύθη, αλλά ήταν και πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί υπήρχαν και άλλα αιτήματα, ενώ αυτή τη φορά μπορούμε να το εξετάσουμε κάθε αυτό. Όπως είπε ο εισηγητής, το Κοινοβούλιο κατάφερε να μην προδικάζει η συμφωνία αυτή τη διαπραγμάτευση για το 2013, τον προϋπολογισμό, δεν προδικάζει δηλαδή πού ακριβώς θα γίνει η ανακατανομή. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο περιθώριο λοιπόν. Όταν χρειαστεί εν καιρό το δέοντι και εν ευθέτω χρόνο θα τα κανονίσουμε. Ούτε θα επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις για το 12, τελείωσαν και αυτές. Και συμφωνούμε ότι δεν θα γίνει καινούργια αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών για αυτό το θέμα μέχρι να λήξει το ισχύον πλαίσιο. Λοιπόν, η Κάρλα, ο Κάρλ με συγχωρείτε, πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εξαιρετικό μας εισηγητή, γιατί η λύση που προτείνει είναι όντως η καλύτερη δυνατή. Κάρλα ιδιαίτερα για το πρόγραμμα για την έρευνα και μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα ζητήσαμε για τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δέχομαι την πρόταση. Δεν υπάρχει εναλλακτική καλύτερη λύση. Ευχαριστώ. Κύριο Σαρτπού. Ευχαριστώ τον εισηγητή κύριε Πρόεδρε. Μας ανέφερε διάφορες ερμηνείες των νομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Ήδη ρωτήσαμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν και τι μας είπαν, ότι με βάση τις συνθήκες επιβάλλεται η ομοφωνία στο Συμβούλιο. Ρωτώ λοιπόν τον εισηγητή, στο Β αναφέρει τριμερή διάλογο του τέλους Δεκεμβρίου 12. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό. Θα γίνει λόγος και τότε για ομοφωνία στο Συμβούλιο τουλάχιστον ή υπάρχουν επιτρέπονται διαφωνίες. Μπορώ να σας απαντήσω αμέσως. Εξορισμού ένας τριμερής διάλογος είναι διαπραγμάτευση μεταξύ εκπροσώπων των τριών θεσμικών οργάνων των δύο πλευρών της αρχής του προϋπολογισμού και της Κομισιόν ως διαμεσολαβητή κατά κάποιον τρόπο. Η Προεδρία της κάθε αντιπροσωπείας του κάθε οργάνου δηλαδή ξέρει ακριβώς ποια είναι η διαπραγματευτική εντολή που διαθέτει. Μας δώσατε διαπραγματευτική εντολή και τα αποτελέσματα θα κρίνεται στην ψηφοφορία για να δείτε αν διαπραγματευτήκαμε καλά. Τα ίδια και ισχύουν και για την Πολωνική Προεδρία. Για την αναθεώρηση του πολιετούς πλαισίου στο Συμβούλιο απαιτείται ομοφωνία. Στο Κοινοβούλιο όμως απλή πλειοψηφία στην Επιτροπή μας και ενισχυμένη στην Ολομέλεια. Κυρία Χέρτσογκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς στην Επιτροπή Βιομηχανίας παρακολουθήσαμε από κοντά το θέμα και θα θέλαμε τα φετινά αποτελέσματα να επαναληφθούν και του χρόνου. Δηλαδή αναφέρομαι για την νίκη η οποία είναι η διατήρηση του προγράμματος πλαισίου 7 και θα θέλαμε να διατηρηθεί να συνεχιστεί και το 13. Δηλαδή και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο και ανάπτυξη και έρευνα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ο κύριος Αρτών... Α, όχι. Ο Ράιμερ θέλει να απαντήσει. Ο Ράιμερ. Κοιτάξτε, το υπενήχθη προηγουμένως, ε, γιατί ε, σας προτείνουμε αυτό το νέο εδάφιο, το Δέλτα κατά την προσαρμογή της ε, θεσμικής ε, συμφωνίας με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πράγματι προκύπτει διαφορετική νομική ερμηνεία από τις υπηρεσίες ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αναθεώρησης του 0,03 του ΑΕΠ. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και η συνέχιση της ε, πολιτικής συμφωνίας. Κατά το παρελθόν είπαμε ότι ε, για μία αναθεώρηση 0,03 το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και πιο πολύ βέβαια με ομοφωνία. Έρχεται τώρα το πρωτογενές δίκαιο ε, το οποίο θίγει από ένα κράτος μέλος και εκεί ορίζεται η ομοφωνία στο δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά ορίζεται επίσης και η μετάβαση σε πλειοψηφικές αποφάσεις. Ε, τώρα, τίθεται το εξής θέμα. Κατά πόσον ισχύει αυτόματα το πρωτογενές ε, δίκαιο ε, και κατά πόσον η δήλωση ενός κράτους μέλους μπορεί να θέσει εκτός ισχύω μία συμφωνία. Εγώ έχω εδώ πάρα πολλές αμφιβολίες. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές νομικές ερμηνείες και η πλευρά του Συμβουλίου είπε ότι ανεξάρτητα με τι θα προκύψει στο μέλλον ε, θα προχωράμε μόνο με ομοφωνία. Ακόμα δηλαδή και το να πάει κανείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα ωφελήσει τίποτα γιατί το Συμβούλιο δεσμεύτηκε μονομερός. Εγώ λοιπόν ε, περιμένω ε, κάποια προγράμματα για τα οποία τα κράτη-μέλη ζήτησαν την ομοφωνία και κάποια εξ αυτών θα βρεθούν σε απελπισία γιατί κάποια άλλα κρατημέλη θα απαιτήσουν αυτήν την ομοφωνία. Κοιτάξτε, η ομοφωνία καταστρέφει την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επιτρέπει να γίνουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ε, ε, με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Γι' αυτό λοιπόν αυτό θέλουμε να αναφέρουμε σε αυτή την παράγραφο. Πράγματι και νομίζω αυτό το είδαμε και στην ε, διαδικασία του προπολογισμού Λόγω αυτής της ε, κατάστασης ε, παρότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση στο Συμβούλιο, ουσιαστικές πολιτικές διαπραγματεύσεις δεν λαμβάνουν χώρα. Απλά οι περισσότεροι στο Συμβούλιο ενδιαφέρονται για κάποιους αριθμούς και οι υπόλοιποι αδιαφορούν. Νομίζω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εδώ κάθε λόγο να προβάλλει τις ευαισθησίες του, ε, κυρίως για το πρόγραμμα ITER, ε, το οποίο ε, μας κόστισε πάρα πολύ χρόνο, αλλά και μεγάλη διασπάθηση ανθρώπινων πόρων. Σας ικανοποιεί η απάντηση. Θέλετε το λόγο. Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Τέθηκε λοιπόν το θέμα στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο για να υπάρξει και η σωστή νομική συμβουλή ε, που θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθούμε και στην νομική υπηρεσία και η Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, επιβεβαίωσαν νομικές τους υπηρεσίες. Κατά τη συνδιαλλαγή του Δεκεμβρίου δεν ξέρω τι θα πει η Πολωνία. Μα δεν είναι αυτό το θέμα, λέει ο Πρόεδρος. Οι νομικές γνωμοδοτήσεις ε, δόθηκαν πριν από ένα χρόνο. Πάει αυτό. Τώρα τι χρειάζεται για να επικυρωθεί και να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Πρέπει να υπάρξει ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το Συμβούλιο πρέπει να θεωρήσει ότι χρειάζεται ομοφωνία. Εάν έχουμε την ειδική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, αν το Συμβούλιο ομόφωνα λάβει απόφαση, εντάξει, λαμβάνει απόφαση. Αν όχι, θα θεωρηθεί ότι το Συμβούλιο δεν συμφωνεί. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο. Εκεί έτσι τίθεται το θέμα, γιατί το νομικό ζήτημα έχει κλείσει, η νομική συζήτηση έχει ολοκληρωθεί. Λύγει το 2013 το δημοσιονομικό πλαίσιο και ξεκινάμε με το νέο, με μια νομική βάση την οποία αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Ράιμερ. Κοιτάξτε, και εγώ το λέω με απόλυτη σαφήνεια. Όχι μόνο το Συμβούλιο ε, θα πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του ε, όταν υπάρχουν διαπραγματεύσει. Αν το Συμβούλιο επέμενε τα σημαντικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα ITER, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο, αν αυτά ε, είχαν απορριφθεί και αν εκεί είχε ζητηθεί η βελτίωση, εγώ θα ερχόμουν εδώ σήμερα και θα σας πρότεινα την απόρριψη. Γιατί πράγματι εμείς ε, ο ρόλος μας δεν είναι να βελτιώνουμε τις ελλείψεις, ε, τις ανεπάρκειες του Συμβουλίου και να το στηρίζουμε, κάθε άλλο. Η κυρία Τρούπελ. Ακόμα και αν ο Ράιμερ είπε τώρα στο τέλος ότι το Συμβούλιο μετακινήθηκε λίγο και ότι η πολιτική Προεδρία ήταν επικοδομητική. Εγώ συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις του Ράιμπερ για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το Συμβούλιο, κυρίως απέναντι στο ε, Κοινοβούλιο. Και όλα αυτά δεν αποτελούν αφορμή για να συνδεξούμε για το μέλλον. Είχαμε μια συνάντηση στο Βερολίνο όπου μας είπαν ότι οι κοινέ δηλώσεις μας ή οι συμφωνίες που προκύπτουν ε, λένε αυτό δεν τους ενδιαφέρει καθόλου γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα και στη τελική ανάλυση αυτό μετράει. Αυτό όμως δεν είναι σωστή αντιμετώπιση και συμπεριφορά ανάμεσα στους θεσμούς και με ανησυχεί πάρα πολύ. Όπως είπε και ο Ράιμερ, εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που λένε μας δώσουμε μια ευκαιρία. Εγώ είμαι ένας από εκείνους ε, που λένε ότι ε, θα πρέπει οι πιστώσεις ε, να καθοδηγούνται, να διοχετεύονται μάλλον σε προγράμματα από τα οποία προκύπτουν νέες τεχνολογίες και νέες θέσεις Γιατί αυτό είναι τμήμα της στρατηγικής που ακολουθούμε το υπάρχει αυτή η αναβολή μέχρι και το 2020 και αργότερα, αυτό δεν είναι έξυπνη απόφαση, αλλά σας λέω, ξέρω ποιες είναι και βλέπω ποιες είναι οι πρωτοβουλίες, λυπάμαι πάρα πολύ και τα λαμβάνω όλα υπόψη μου. Ε, και να πω και άλλη μια φορά, οι πράσινοι δεν θα συμφωνήσουν με αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο Ιβάνο Κάλφιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω καταρχάς ότι συγχαίρω τον Ράιμερ για τις διαπραγματεύσεις και για το αποτέλεσμα που επέτυχε. Γιατί γνωρίζουμε ότι αρχικά η θέση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Με τα 360 εκατομμύρια το 2013 θα έχουμε το πρόβλημα, νομίζω. Πρέπει να αποφασίσουμε από τώρα τι θα γίνει τότε και πριν ξεκινήσει η διαδικασία για το 2013 να μην αναλάβουμε κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Νομίζω ότι είχαμε πει ότι τα 360 εκατομμύρια θα αποφασιστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας για το 2013. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα είναι πρόταση της Κομισιόν, αλλά πρέπει να δούμε πώς οργανώνεται και από πού προέρχεται αυτή η χρηματοδότηση γιατί θα ήθελα για μια ακόμη φορά να επαναλάβω τη θέση της δικής μας πολιτικής ομάδας, ότι δηλαδή δεν είναι καλή ιδέα να επαναναπτύξουμε ποσά τα οποία έχουν αναδεθεί στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο σε κοινοπραξίες. Χαίρομαι που δεν θα γίνει αυτό τώρα, αλλά πρέπει τελικά να το ξανασυζητήσουμε. Για τον προπολογισμό του 2013, επαναλαμβάνω. Τουλάχιστον για δύο χρόνια είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα για το ίτερ. Μετά μπαίνουμε στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και εκεί δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Merci, mon cher Bien. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ η συζήτηση. Σας προτείνω να περάσουμε στις ψηφοφορίες τώρα. Για να τηρήσουμε λίγο και το χρονοδιάγραμμα. Θα ψηφίσουμε για το ίτερ και για τις λοιπές εκθέσεις και μετά θα ασχοληθούμε με τα άλλα σημεία της μερίσιας διάταξης που δεν έχουμε εξετάσει ακόμη. Λοιπόν, για το ίτερ σας προτείνω να ψηφίσουμε unblock συνολικά για την έκθεση Ρέμερ Μπέγκε, όπως τροποποιείται με δύο προφορικές τροπολογίες. Τις έχετε λάβει αυτές τις ε, προφορικές τροπολογίες, έτσι. Συμφωνείτε να ψηφίσουμε unblock. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιοι είναι κατά. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Nine, nine, τι ο nine, nine. Είναι, είναι υπέρ. Ναι, ναι, μα το... Δεν τη μετράω την Ίνγε Την Ίνγε συνηθίσαμε, δεν την μετράμε στην Επιτροπή Προεπολογισμών. Αστείευομαι, αστείευομαι. Είναι δύο εδώ και δύο από εκεί. Λοιπόν, αποχές. Δεν υπάρχει κάποιος. Σας ευχαριστώ λοιπόν, μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης. Τώρα, συγχαίρω φυσικά τον εισηγητή και τώρα. Την επόμενη Τρίτη στην Ολομέλεια ψηφίζουμε μετάφραση σε όλες τις γλώσσες μεθαύριο. Άρα είμαστε μέσα στις προθεσμίες για να μπορέσουμε πράγματι να ψηφίσουμε την επόμενη Τρίτη. Προτείνω τώρα να περάσουμε σε μια άλλη έκθεση του Ράιμερ Μπέγκε δηλαδή την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την Ισπανία και για την Ιταλία. Μία ψηφοφορία μόνο. Ναι. Απλά να σας πω το εξής. Υπάρχει ένα σφάλμα, τεχνικό πρόβλημα. Δυστυχώς παρισέφρισε ένα σφάλμα στην έκθεση για την πρόταση ψηφίσματος. Παράγραφος 3 συγκεκριμένα αυτόματη παράγραφος ε, την οποία βάζουμε σε κάποιες ε, περιπτώσεις. Εδώ δεν ε, θα έπρεπε να είναι η παράγραφος 3, άρα δεν θα ψηφίσουμε για την παράγραφο 3. Η δεν αφορά την παράγραφο 3. Ποιοι είναι υπέρ της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Ψήφισε και ο εισηγητής πριν φύγει. Κατά ποιοι είναι. Αχτονκ. Αποχές. Βέρτμαν. Μία αποχή δηλαδή. Άρα εγκρίνεται και συγχαίρω τον εισηγητή. Τώρα, για τον διορθωτικό προπολογισμό 7 του 2011. Μία ψηφοφορία για την έκθεση στη Συντόνια που δεν είναι εδώ. Είναι υπέρ βέβαια συγκήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Κατά. Ένας. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, για το πρωτόκολλο με τη Δημοκρατία της Γνέας Μπισάου για την Αλία. Το συζητήσαμε δύο μακρόν. Δύο φορές συγκεκριμένα το συζητήσαμε. Δύο ψηφοφορίες έχουμε. Πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε την έγκριση του πρωτοκόλου, του αλληλευτικού πρωτοκόλου. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ένας. Αποχές. Ουδής. Άρα εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ένας. Αποχές, καμία. Άρα το ίδιο, όπως και στην προηγούμενη. Για την έκθεση ματέρα τώρα. Ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. η κινητοποίησή του για τον Τρεντίνο, Άλτο Άντιτζε και τον Νότιο Τυρόλο. Δύο εκθέσεις είναι διαφορετικές. Λοιπόν, έχετε τις λίστες. Έχουμε κάποιες τροπολογίες. 1-7. Λοιπόν, τροπολογία 3 των φιλελευθέρων. Υπέρ είναι η συγκήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. σοσιαλιστές είναι κατά. Μάλιστα. 3-4-5. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 των ίδιων συντακτών. Η συγκέντρια είναι αντίθετη όμως εδώ. Υπέρ. Η φιλελεύθερη κυρία Βέρτμαν. Κατά. Πλειοψηφία από τη βλέπω. Αποχές απορρίπτεται. Πέντε Βέρτμαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Έξι Φιλελευθέρων. Η συγκέντρια είναι κατά. Ψήφι υπέρ. Αχά, αχά, αχά, λέει ο πρόεδρος. Ποιοι είναι κατά. Πρέπει να μετρήσουμε. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της 6 παρακαλώ. Ξανασηκώστε τα χέρια. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ποιοι είναι κατά παρακαλώ. Εγκρίνεται η 6. 7. Ίδιων συντακτών. Συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Οι σοσιαλιστές εν κατά αποχές εγκρίνεται. Πολύ διασκεδαστικό. Οι ίδιοι συντάκτες υποστηρίζονται ή δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την τροπολογία. Επτά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Οι ίδιοι πάλι εγκρίνεται. Οι δύο Βέρτμαν υπέρ. Πολύ. Κατά. Η φιλελεύθερη είναι κατά. Μάλιστα. 4-5-6. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Δύο ψήφοι κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Άρα. Α, έχουμε. Έχουμε. Ο Τζέιμ. Ο Τζέιμ απέχει. Μάλιστα. Εγκρίνεται λοιπόν. Τώρα έχουμε τα εμβάσματα τώρα, τις μεταφορές πιστώσεων. Θα ξεκινήσουμε από τα άλλα θεσμικά όργανα, περιμένοντας τον συγκητή για την Επιτροπή να έρθει στην αίθουσα. Η Χέλγα λοιπόν τώρα να μας, παρα... Ε, να μας εκθέσει τα δικά της εμβάσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω εδώ υποθέσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και προσφυγές που αφορούν μεταφορές και τις λεγόμενες σκουπιστικές επιχειρήσεις. Mopping up operations. Το συνολικό ποσό είναι 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Είχα εκφράσει αμφιβολίες για αυτή τη μεταφορά και την περασμένη φορά γιατί λόγω της δύσκολης κατάστασης πολλών χωρών μελών καλύτερο θα ήταν να επιστραφεί το ποσό στα κράτη-μέλη. Αλλά φαίνεται ότι δεν το χρειάζονται οι χώρες. Δεν το απαιτούν. Και γι' αυτό συστήνω άντε να το εγκρίνουμε. Το Άψογα ευχαριστούμε. Ποιος είναι υπέρ αυτής της μεταφοράς που προτείνει η συγκήτρια. Ευχαριστούμε. Τις τρεις μεταφορές, τρεις μεταφορές και όλες μαζί. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνονται. Τώρα κυρία εισηγήτρια μου. Το EAS επίσης θα ήθελε τα χρησιμοποιεί τα κονδύλια ύψους ενός εκατομμυρίου να χρησιμοποιηθούν για να του επαναδιατεθούν για θέματα προσωπικού. Εγώ δεν είμαι κατά, δεν είμαι κατά. Για την υπηρεσία λοιπόν εξωτερικών δράσεων. Ποιος είναι υπέρ, κατά, ένα αποχές, καμία. Η μεταφορά εγκρίνεται, ευχαριστώ. Τώρα κυρία εισηγήτρια, για τα κτίρια, ξέρετε ότι έχουμε πρόβλημα με το κτίριο εκεί στο Στρασβούργο και το Μοντουαγέλα. Είπαμε την επόμενη εβδομάδα να το συζητήσουμε τη Δευτέρα, εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα λοιπόν. Τελευταία μεταφορά για το Κοινοβούλιο αφορά το topping up 2,3 εκατομμυρίων από προηγούμενο προϋπολογισμό με δικαιολόγηση ότι πρέπει να καλυφθούν κενά στις πληροφορικές δομές. Και να προβλεφθούν ανάγκες του 12 καθώς και προγράμματα υποδομών. μέσω της συνέχισης της χρησιμοποίησης εξωτερικών υπαλλήλων. Στους όλους τους τόπους εργασίας και συστήνω έγκριση και αυτής της μεταφαράς. Α, μάλιστα, η γάμα 8 δηλαδή, ο Τζέιμς. Επειδή δεν τα ξέρω όλα κύριε Πρόεδρε, τι είναι το κέντρο δεδομένων των Βρυξελών που άκουσα. Είναι εξωτερική υπηρεσία, είναι εσωτερική, τι είναι. Κυρία εισηγήτρια, αν επαναλάβει γιατί δεν άκουσα. Διάβασα εδώ την εξήγηση τη δικαιολόγηση της μεταφοράς και αναρωτιέμαι τι είναι Brussels Data Center. Είναι μια εσωτερική υπηρεσία, εξωτερική, ποιος το διαχειρίζεται κλπ. Ίσως έχετε κάποια εξήγηση εσείς. Κάποιος από τη διοίκηση είναι εδώ να μας απαντήσει γιατί εγώ δεν ξέρω. Ναι, ναι, υπάρχει από την υπηρεσία κάποιο. Κύριε Διευθυντά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι εγκαταστάσεις που έχουμε εκτός των κτηρίων ως backup των συστημάτων μας. Και αυτή τη στιγμή αγοράζουμε μηχανήματα αυτού του νέου κέντρου δεδομένων για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας. Εκτός και με εκτός και των συνήθων υπαλλήλων, ή με τους συνήθους υπαλλήλους, αλλά εκτός. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ψηφίζουμε αυτή τη μεταφορά γάμα 8 υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Καμία. Εγκρίνεται λοιπόν και αυτή. Δεν έχετε άλλες μεταφορές, ΕΛΓΑ. Ωραία γιατί για τα κτίρια είπαμε θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ο άλλος εισηγητής, η Σιδονία δηλαδή, για τις μεταφορές που αφορούν τον προπολογισμό της Κομισιόν. Ορίστε κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχει μια σειρά μεταφορών και εδώ, παρόμοιων με τις προηγούμενες δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί όμως όλες γιατί κάθε μία είναι διαφορετική περίπτωση. Να τις δούμε μία-μία λοιπόν. Η πρώτη αφορά την κινητοποίηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης αλλά επειδή ήρθα καθυστερημένη δεν ξέρω αν συζητήσατε αυτή την έκθεση αν ναι Πάντως εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο να αρνηθούμε την μεταφορά αυτήν. Ευχαριστώ. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς 28 λοιπόν. Μάλιστα κατά. Αποχές. Ευχαριστώ εγκρίνεται. Ή 48 τώρα. Η μεταφορά αυτή αφορά τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στην... στη συνδιαλλαγή και αφορά 69,3 εκατομμύρια για την υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θυμάστε τα μέτρα για την βανάνα. Είχαμε πει τότε ότι η συνδιαλλαγή που έγινε με όλα τα όργανα ήταν να μεταφερθούν μερικά από τα ποσά εκείνα που περίσευαν. Αυτό συμφωνεί και με τη συμφωνία που είχαμε κάνει στην για την Ολομέλεια. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ναι, συμφωνία λοιπόν για τα ΕΣ παράγωγες πράξεις, μάλιστα είναι για την βανάνα όπως είπαμε. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής, στο κατά. Αποχές, μία ψήφος κατά. Η μεταφορά 50. Η μεταφορά αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι έχει υπάρξει καθυστέρηση ορισμένων προγραμμάτων στην θέση συνεργασία με τρίτες χώρες για θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Και ο λόγος της μεταφοράς είναι για να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια αυτά υπό το πλαίσιο του DCI. Δεν έχω αντίρρηση ούτε εδώ. Μάλιστα, ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς 50, κατά, ευχαριστώ αποχές, εγκρίνεται η 51. Η μεταφορά αυτή συνδέεται με μια ρύθμιση στη Γενική Διεύθυνση Περίφ δεν βλέπω καμία κανένα αντίρρηση. Μάλιστα, ποιο είναι υπέρ τη μεταφορά 51. Μάλιστα, κατά. Ευχαριστώ, αποχέ. Εγκρίνεται η 52. Η μεταφορά αυτή πρέπει να εξηγηθεί λίγο περισσότερο. Θα ήθελα να σας δώσω μερικές πληροφορίες. η μεταφορά αυτή συνδέεται πάλι σε μια συμφωνία στη συνδιαλλαγή. Ίσως θυμάστε ότι η Κομισιόν είχε ζητήσει 550 εκατομμύρια στη συνδιαλλαγή δεχτήκαμε 200 το 11 και βέβαια υπάρχουν και άλλες ανάγκες που δεν καλύπτονται από αυτή την απόφαση. Γι' αυτό έχουμε αυτή την πρόταση μεταφοράς 52. 600 εκατομμύρια. Και στο φάκελό σας βλέπετε ότι χρειάστηκε να συνδυαστούν πολλές θέσεις μαζί για να καταλήξουμε σε αυτό το ποσό είναι οι πληρωμές που χρειάζονται για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τις κοίταξα όλες αυτές τις θέσεις για να δω ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της εφαρμογής αυτής της πρότασης και από πού προέρχονται τα χρήματα. Και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αναβολή πληρωμών μέχρι τον Ιανουάριο απλώς. Η Κομισιόν δηλαδή ταύτισε τα προγράμματα της θέσης του προϋπολογισμού όπου μπορούν να αναβληθούν οι πληρωμές μέχρι τον Ιανουάριο. Εγώ δεν είμαι όπως ξέρετε υπέρ τέτοιων λύσεων αλλά αφού προκύπτει από συμπεφωνημένα στη συνδιαλλαγή πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα θα είναι περαιτέρω δημοσιονομική πίεση το 12 αλλά δεν είναι το δικό μου θέμα δεν μπορώ να μιλήσω για το 12, αλλά σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό και το 12. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Να σας πω μερικές από τις λεπτομέρειες των θέσεων. Μερικές αφορούν το άσυλο, την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης και θα πληρωθούν τον Ιανουάριο. Είχαν προβλεφθεί για τον Ιανουάριο του 2011. Είχα ζητήσει από την Κομισιόν να μου πει πώς επιλέγουν τι αναβάλλεται και τι όχι. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η ερώτηση. για οποιονδήποτε πληρωτή και μου είπαν ότι τουλάχιστον για τα διαρθρωτικά προγράμματα πληρώνουν όποιον έρθει πρώτος, όποιος το ζητήσει πρώτος, όποιος υποβάλλει το λογαριασμό πρώτος. Γι' αυτό μερικά προγράμματα πληρώθηκαν από τις αρχές του 11 και άλλα όχι. Αν έχετε απορίες, η Κομισιόν να σας απαντήσει. Εμένα πάντως μου είπαν ότι αυτή η καθυστέρηση στις πληρωμές οφείλεται σε αυτό που σας είπα. Μάλιστα, ευχαριστούμε κυρία Σιδανία. Πράγματι, αυτά οφείλονται στη συμφωνία μας, στη συνδιαλλαγή και στην ψηφοφορία που κάναμε στην περασμένη Αλαμέλεια. Ο κύριος Χάρτουγκ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με αυτές τις προτάσεις που ακούσαμε Ουσιαστικά πρόκειται για κάποια νούμερα για του χρόνου και θα δούμε αν μπορούν να πληρωθούν ή όχι μετά. Μα δεν μπορώ να πω ότι είναι και η πιο ωραία προσέγγιση αυτή. Θα ήθελα να ζητήσω κάποια σχόλια από την Κομισιόν για τις επιπτώσεις. Τα 550 εκατομμύρια, από ό,τι θυμάμαι, ήταν χαμηλότερο από το αρχικό νούμερο που είχαμε εκτιμήσει εμείς, που ήταν το διπλάσιο περίπου. Και τώρα πέσαμε στα 550, 200 και θα κάνουμε αυτή τη μεταφορά. Αυτές είναι ανάγκες του Ευρωπαϊκού Ταμείου και άλλων τομέων προτεραιότητας. Τι ε, πιέσεις παραπάνω θα ασκήσει αυτό στον προπολογισμό. Έχουμε ένα πιο συνολικό νούμερο. Δηλαδή η Κομισιόν μπορεί να μας εξηγήσει τελικά τι σημαίνει αυτό για την υλοποίηση των προγραμμάτων και για την επιπλέον πίεση στον προπολογισμό του 2012. Πρόεδρος, πράγματι μιλάμε για backloading ε, μεταφορά στην αρχή της επόμενης χρονιάς για πληρωμές που δεν μπορούμε να κάνουμε φέτος. Αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον θα απαντήσει η Κομισιόν, η Χέλκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι και εγώ σε αυτό γιατί όταν διάβασα τα έγγραφα και άκουσα αυτά που λέει η Συντονία δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες αν επανάπτυξη των 600 ε, εκατομμυρίων. Αυτό που οφείλεται, καθυστερήσατε να πληρώσετε το ποσό, αυτό που λέει ο πρόεδρος Λαμασούρ, ή δεν δαπανήθηκαν οι πόροι για οποιοδήποτε λόγο. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση για να το καταλάβω. Και στη διάρκεια της συνδιαλλαγής είχαμε πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο η Κομισιόν μπορεί να βρει τα χρήματα μπορούν, δεν μπορούν. Κάτι που θα αποδείξει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι. Άρα θα μπορούσε αυτό να τερμινεύσει κανείς, μην πληρώσετε το 2011, αλλά αναβάλλετε την πληρωμή για το 2012. Είναι σημαντική πληροφορία. Πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται ακριβώς και θέλω μια διευκρίνηση. Ε, Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ο πρόσωπος Κομισιόν παρακαλώ. Πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει περισσότερες πληρώμες από αυτές που επιτρέπει ο διορθωτικός προϋπολογισμός 6 ε, ε, Εκεί είχαμε ένα χαμηλότερο ποσό πληρωμών. Εμεί προσπαθούμε να εξοπλίσουμε κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις διαθέσιμες πληρωμέ, για να καλύψουμε τις έκτακτες ε, ανάγκες και αιτήματα που εκτιμώνται σε 1,5 δι και για το κοινωνικό ταμείο και για τα άλλα. 450 εκατομμύρια περίπου <laughs> τα βρήκαμε το διορθωτικό προπολογισμό 6. Με αυτή τη μεταφορά πίστοσης, γύρω στα 600 εκατομμύρια πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Ελληνικό Ταμείο. Και έχουμε μία εκκρεμότητα ακόμη, γύρω στα 450 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη μεταφορά, 600 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι αυτά τα ποσά. Μιλάμε για πιστώσεις πληρωμών αφού πέρασαν από όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Πρόκειται για πληρώμες που είτε δεν θα χρησιμοποιούσαν μέχρι το τέλος του έτους, ή υπήρχε κίνδυνος να μην χρησιμοποιούν μέχρι το τέλος του έτους. Εξού και η μεταφορά πίστοσης που προτείνει να χρησιμοποιηθούν για έκτακτα αιτήματα που εκκρεμούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τώρα, τα αναπομένοντα 450 εκατομμύρια τώρα. Τι θα γίνει με αυτά. Συνήθως στην υλοποίηση της για το Κοινωνικό Ταμείο, ε, περιφερειακό, ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχουμε την υλοποίηση μέχρι το τέλος του χρόνου. Εάν στο τέλος του χρόνου κάποιες από τις αναμενόμενες πληρωμές δεν έχουν γίνει ιδίω για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Κομισιόν θα προσπαθήσει ό,τι υπόλοιμα υπάρχει, ό,τι υπόλοιπο υπάρχει να το χρησιμοποιήσει για να, χρησιμοποιεί, για να καλύψει μέρος ε, των αναγκών του ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλησης, κυρίως. Και κάποιες από τις του Κοινωνικού Ταμείου επίσης θα καλυφθούν με αυτήν την εκ νέου ανάπτυξη. Έχουμε την ε, εξουσιοδότηση να το κάνουμε αυτό εσωτερικά στην Κομισιόν. Μέρος των αργών δεν θα καλυφθούν. Εξού και θα χρειαστούν μεγαλύτερες ε, πιστώσεις πληρωμών για το 2012. Και θα υπάρχει πρόβλημα με άλλες ανάγκες. Θα ανταγωνίζονται οι μεν τις δε. Και ίσως πράγματι προκύψουν δυσκολίες γύρω στα τέλη του επόμενου έτου. Θα έχουμε ανεπάρκεια στις πιστός πληρωμέ. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε λοιπόν ε, την υλοποίηση και να μπορέσουμε εκ των προτέρων να εντοπίσουμε πιθανές ανάγκες που δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν. Αυτό θα το δούμε του χρόνου. Merci, Geran. Geran Συγγνώμη, αλλά είχα ξεχάσει κάτι. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω ακόμη. Έχουμε κάποιες γραμμές προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά θα ήθελα μία ακόμη γραμμή για την ε, Παλαιστίνη. Στην συνδιαλλαγή κάναμε ένα front loading ε, των δεσμεύσεων για το 2011, αλλά υπάρχει και τεράστια ανάγκη για πληρωμές. Μα είπαν από την Άμρα πριν από κάποιες ημέρες ότι υπάρχει θέμα με την πληρωμή μισθών ε, των εκπαιδευτικών, ε, των δασκάλων για του των Δεν μπορούν να καταβληθούν το Δεκέμβριο. Άρα θα έλεγα ε, ότι έπρεπε να υπάρχει αυτή η γραμμή για την Παλαιστίνη που δεν υπάρχει. Μπορεί να το σχολιάσει αυτό η Κομισιόν. yes, as far as the... Σε ό,τι αφορά τη βοήθεια προς την Παλαιστίνη, δεν ε, μας ενημέρωσαν ε, ότι υπήρχε πρόβλημα στις πληρωμέ. Γιατί είναι σε ένα άλλο κονδύλιο. Οι σχετικέ πληρωμές δεν ε, γνωρίζω να υπάρχει πρόβλημα στις πληρωμέ για το 2011. Μάλιστα, αν κατάλαβα καλά την απάντησή σας, λέει ο Πρόεδρος, μπορείτε να, εξασφαλί... να τον Γκέραν Φέρμ ότι τα χρήματα τα οποία προβλέπονταν στην συμφωνία που επιτέχθηκε στη συνδιαλλαγή θα, διατεθούν. Δεν είναι θέμα για τη συγκεκριμένη μεταφορά. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό για τη συγκεκριμένη μεταφορά. Ωραία, ο κύριος Χάρτονγκ. Ναι, έχω μια ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά. Ο προϋπολογισμός του 2012 έχει ε, ξεπεραστεί, αν μπορώ να το πω έτσι, πριν καν ξεκινήσει ο χρόνος. Δηλαδή έχουμε ήδη εξαντλήσει τα περθ... Όχι, όχι, λέει ο πρόεδρος, όχι. Καθυστερούμε για το 2012 κάποιες δαπάνες που θα έπρεπε να είχαν γίνει το 2011. Τις αναβάλουμε για το 2012. Τώρα τι θα γίνει σε όλο το 2012 θα το δούμε. Μετά από όλες αυτές τις ε, επεξηγήσεις ε, η συγκήτρια ε, δίνει θετική, δίνει το πράσινο φως για αυτή την μεταφορά πίστοσης. Ναι, είμαι υπέρ αυτής της μεταφοράς αλλά να απαντήσω ε, δύο συγκεκριμένα ερωτήματα της Χέλγα Τρούπελ και του κυρίου Χάρτονγκ για την κυρία Τρούπελ. Πράγματι, υπάρχει ένα μείγμα καθυστερήσεων και, όχι επαρκούς, και ανεπαρκούς υλοποίησης, under ε, exploitation. Σωστά το είπατε και το επισημάνατε αυτό. Στην επεξήγηση που λάβαμε στο αρχικό DEC 53 φαίνεται ότι υπάρχει ανεπαρκή υλοποίηση, under implementation, συγγνώμη, και όχι exploitation, under implementation. Δυστυχώς ε, μιλάμε για μεγάλο ποσό. Θα το δείτε σε κάθε γραμμή, εκεί που δεν υπήρξε πλήρης ε, υλοποίηση. Μη εκμεταλλευτήσεις πιστώσεις τις λέμε. Αλλά δεν είναι κάτι επίμαχο για μένα. Το τόνισα και είπα όμως ότι τι είναι αυτό που με προβληματίζει. Πάντοτε με προβληματίζουν οι αναβόλες στις πληρωμές. Και αυτό έχει να κάνει και με αυτό που είπε και ο κύριος Χάρτονγκ. Είπατε είναι αυτό καλή ε, κατάρτιση προπολογισμού, good budgeting. Όχι, δεν είναι. Αλλά μιλάμε για πιστώσεις πληρωμών από τα κράτη-μέλη που δεν ήθελαν καν ε, να έχουμε φρέσκο χρήμα 200 εκατομμύρια. Και καθόμαστε όλο το βράδυ και περιμέναμε μέχρι να καταλάβουν τελικά τα κράτη-μέλη έπρεπε να προσθέσουν ε, επιπλέον πιστώσεις πληρωμών για το 2011. Άρα, όπως σας είπα, πρέπει να επανέλθουμε του χρόνου σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες υποχρεώσεις και προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά απροθυμία από τα κράτη-μέλη να πληρώσουν. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά οφείλεται στο ότι δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να δώσουν ε, την απαιτούμενη χρηματοδότηση για το επίπεδο των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. Ε, πολύ σύντομα να σας πω το εξής. Ε, το κοινωνικό ταμείο είναι εκείνο που καταβάλλονται τα χρήματα γιατί έχει να κάνει κυρίως με ήπια προγράμματα. Γι' αυτό το λόγο έχει καλύτερη απροφητικότητα από το Περιφερειακό Ταμείο που και αυτό έχει κάποια σχέση με την περιφερειακή υποδομή. Νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε την πρόταση του εισηγητή γιατί αν δεν στηρίξουμε αυτό το ταμείο τότε ε, καταλαβαίνετε θα υπάρξει πρόβλημα. Βέβαια υπήρξε μία περικοπή κατά ένα εκατομμύριο στις ε, πληρωμές, όχι στο κοινωνικό ταμείο, αλλά κυρίως ε, όσον αφορά τα κονδύλια που διατίθενται στις ε, προηγμένες χώρες. Εμείς δεν προβήκαμε σε καμία αλλαγή και είχα το λόγο ο ε, τροποποιητικός προπολογισμός ξεκινάει από τον Ιανουάριο ακόμα και αυτή την αναβολή, με αυτήν την αναβολή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα στο τέλο του έτου δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να μην στρίψουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά από τι παρατηρήσει και επεξηγήσει αυτέ που ήταν πολύ χρήσιμε, προτείνεται να εγκρίνουμε τη μεταφορά αυτή. ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Στο αποχές. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Τι μένει τώρα η 53 κυρία εισηγήτρια. Η μεταφορά 53 αφορά τους ισολογισμούς και τις ψηφισμούς, δηλαδή ξέρετε και είναι στις θέσεις του προϋπολογισμού που ε, δεν έχουν ακόμη κλείσει μέχρι τώρα μερικά κράτη-μέλη πρέπει να ζητήσουν αύξηση κατά 16 εκατομμύρια, δηλαδή σύνολο 320. Από διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού προβλέπονται οι αυξήσεις αυτές. Μία από αγροτικές δαπάνες, η υψηλότερη αφορά την αποθήκευση δημητουριακών για τις παρεμβάσεις και το γάλα σε σκόνη. Όλα αυτά ισοδυναμούν με τις προβλεπόμενες ε, πιστώσεις. Δεν υπάρχει δυσκολία ούτε σε αυτή τη μεταφορά. Σας ευχαριστώ. Ναι, είναι ο συμψηφισμός μάλιστα που γίνεται παραδοσιακά στη Γεωργία στο τέλος του έτους. Ποιος είναι υπέρ, ευχαριστώ κατά, Εποχές, Ευχαριστώ. Έληξαν οι ψυχοφθορίες Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Τι έχουμε τώρα, δύο σημεία για ανταλλαγή απόψεων, σύντομη όμως σύντομη. Πρώτον το 8, η γνωμοδότηση της κυρίας Βέρτμαν δηλαδή, για το καθεστώς του δικαστηρίου. Ορίστε κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ τον Μάρτιο αυτού του έτου, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προέβησε διάφορες αλλαγές του καταστατικού του. Σύμφωνα λοιπόν με τη συνθήκη της Λισαβόνας αυτές οι τροποποιήσεις ε, πρέπει να εγκριθούν και από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προτινόμενες αλλαγές αφορούν τα τρία δικαστήρια, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Δικαστήριο για τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Εδώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαστήριο επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Δύο προτάσεις αφορούν αλλαγές προσωπικού, οι οποίες αλλαγές ε, προφανώς ε, συνεπάγονται υψηλότερο κόστος και έχουν σημασία για τον προϋπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προτείνει και την θέση του ε, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αυτό εξηγείται με το ότι πραγματικά ο Πρόεδρος τη διάρκεια όλων των τελευταίων ετών επιβαρύνθηκε τα μάλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κουράστηκε βέβαια, αλλά απλά σημαίνει ότι υπάρχει ε, φόρτος εργασίας ε, και δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήσουν έγκαιρα τουλάχιστον οι υποθέσεις. Ε, έτσι λοιπόν ε, πολλοί αναγκάστηκαν να περιμένουν μέχρι και ένα χρόνο για να ε, διεκπαιρωθεί μια δικογραφία. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Το επιπρόσθετο κόστος περιλαμβάνει ε, τις, ε, τους μισθούς, ε, τις αποζημιώσεις και η δεύτερη αλλαγή που προβλέπεται είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προτείνει ο αριθμός των, των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αυξηθεί στους 12 και επιχειρηματολογεί με το ότι υπάρχει ανισορροπία. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο αριθμός ε, των εκκρεμουσών υποθέσεων αυξάνεται συνεχώς και εδώ λοιπόν ε, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ή αναγκασμένοι να περιμένουν πάρα πολύ και αν δει κανεί ε, τον ε, αριθμό των 300 υποθέσεων που εκκρεμούσαν στο τέλος του 2010, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Φέτος εξετάστηκαν μόνο 25 υποθέσεις. Βλέπω λοιπόν να υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι ο αριθμός των υποθέσεων θα αυξάνεται κατέτος. Για μας αυτό που παίζει βέβαια ρόλο είναι το κόστος. Ε, το πρώτο έτος θα υπάρξει σημαντική αύξηση 13,65 εκατομμύρια θα είναι την δεύτερη χρονιά. Είναι σαφές ότι λόγω της οικονομικής μας κατάστασης και της οικονομικής κρίσης στα κράτη-μέλη ε, Ίσως αυτό ή αυτά τα ποσά να μοιάζουν υπέρογγα, Από την άλλη όμως πρέπει κανείς να έχει κατά νου ότι ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δουλεύει σε ένα ε, χρονικά αποδεκτό πλαίσιο και θεωρώ ότι το να έχουμε ένα ανεποτελεσματικό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό θα προκαλέσει στην κοινωνία ακόμα μεγαλύτερο κόστος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ κρίνω ότι αυτή την ε, αίτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τροποποίηση του κατσατικού του πρέπει να τη δεχτούμε και ε, όσον αφορά την κατάθεση τροπολογιών ε, προβλέπεται η 14η Δεκεμβρίου. Για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είμαι στη διάθεσή σας και νομίζω ότι ε, όπως και την τελευταία φορά πρέπει όλοι να αποφασίσουμε από κοινού βεβαίω και να συζητήσουμε η ψηφοφορία προβλέπεται, η ημερομηνία ψηφοφοριας προβλέπεται 25 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε κύριε Σιγήτρια, ξεκάθαρα ήταν. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια, όχι. Όπως λοιπόν είπε η κυρία Φέρτμαν, έχουμε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για τις 14 Δεκεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Έχουμε προβλέψει να ψηφίσουμε την γνωμοδότησή μας στις 25 Ιανουαρίου, ώστε να μπορεί έγκαιρα η Νομική Επιτροπή να ψηφίσει στις 26 Ιανουαρίου και μετά πάει η έκθεση στην Ολομέλεια. Τελευταίο σημείο στη Μερσία διάταξη τώρα είναι η έκθεση Godmanis. Παριθμόν 9 σημείο τη μερική διάταξη. Ρόλο τη πολιτική συνοχή στι ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιφέρειε. Η Λετωνία μεταξύ αυτών. Ε, because it's very late and I do believe that the people... Είναι πολύ αργά και θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή πόσο δεν θα μακρηγορήσω. Είμαι μέλος Επιτροπής ε, Ρέτζι, όχι τακτικό, όχι πλήρε. Και είμαι και σκιώδη συζητητή για το νέο νομοθετικό πακέτο. Τα έγγραφα δηλαδή που αφορούν τη νέα πολιτική συνοχή. Είμαι ο σκιώδης από την ομάδα μου. Και μόλις αρχίσαμε να συζητάμε αυτά τα έγγραφα στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ρέτζι πρέπει να πω στην Επιτροπή Προπολογισμών για μια ακόμη φορά ότι θα έχουμε πολλές προτάσεις από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΡΕΤΖΙ. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα συμφιλώσουμε τα πράγματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλία για τι ιδιαίτερε απομακρυσμένε περιφέρειε. Μετά θα έχουμε άλλα έγγραφα, καινούρια έγγραφα από, τη γάμα δελτα, από την ε, κύριος Κάλφιν ίσως να είναι αυτός που θα είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά. Και είναι ενδιαφέρουσες προτάσεις. Είναι προτάσεις ότι δηλαδή θα μπορούσε να δίνει εγγύηση σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε εθνικές τράπεζες για να παρέχουν συγχρηματοδότηση για έργα συνοχής σε περίπτωση που εθνικές τράπεζες δεν δίνουν δάνεια για να ξεκινήσουν τα έργα. Είναι σταρπαστικό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Για το ε, έργα οδοπίας, 4,5 δίσε. Για την Ελλάδα. Και θα δοθούν κάποιοι πόροι, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κρατημέλη, κάπως περίεργη η κατάσταση. Από την τα Ρέτζε θα έχουμε κάποιες τέτοιες προτάσεις. Και εκεί εντάστηκε αυτή η έκθεση. Γιατί οι κανονικές συνθήκες αρχίσουν όλοι να λένε ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Δεν ξέρω αν ε, το έχετε μελετήσει στην Επιτροπή σας αρκετά, αλλά έχω ξαναπεί Μιλάμε για τον προπολογισμό 14-20. Εκεί έχουμε ένα παιχνίδι. Τα χρήματα της συνοχής δεν αυξάνονται. Φαίνεται να είναι πιο υψηλά τα ποσά για τον πολύ απλό λόγο ότι η Κομισιόν βάζει 40 δις στη συνοχή και αυξάνεται το ποσό, αλλά στο πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο ήταν εκτός του 1β αυτά τα ποσά. Εάν δείτε προσεκτικά τις προτάσεις συνοχής. Υπάρχουν κάποιες περιφέρειες που μειώνται ε, τα κονδύλια κατά 20%. Αν δείτε τις τιμές είναι συγκρίσιμες. Είναι 203 δις στο Υπάρχουν ε, MMF και μετά θα είναι 162. Γιατί, γιατί δεν υπάρχουν καθόλου πόροι για τις μεταβατικές ε, περιφέρειες. Αν δείτε το phasing out και το phasing in είναι γύρω στα 40 δις. Για τις περιφέρειες που θα πάνε στο πάνω από το 75%. Τι λέω, τι θέλω να πω. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες περιφέρειες όπου η Κομισιόν για το επόμενο πολιτές μεσονομικό πλαίσιο δεν θα αναθέσει χρήματα, δεν θα διαθέσει συγκεκριμένα, θα προβλέψει συγκεκριμένο κονδύλιο. Ήταν 0,99 δις στο τρέχον πλαίσιο και θα είναι 0,92 δις στο επόμενο συγκρίσιμα είναι ε, κοντά, συγκριτικά κοντά. Για ποιες περιοχές μιλάμε, για ποιες περιφέρειες. Μιλάμε για τα Κανάρια, για τη Μαδέρα, για τις Αζόρες, ε, για τα γαλλικά υπερποντια μερίσματα. Δηλαδή για περιοχές μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ξεκάθαρο. Ουσιαστικά όποιος είναι μακριά πρέπει και να έχει μεγαλύτερη στήριξη, αλλά ε, αν το δούμε υπό το πρίσμα της Επιτροπής Περιπολογισμών, Ακόμη και αν πρέπει να συζητήσουμε πρώτα πώς αντιδράμε σε σχέση με το συνολικό πακέτο, ε, τα νομοθετικά αυτά πακέτα που πρέπει να τα περιμένουμε σύντομα από την ΓΔΡ και θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε γι' αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο ένα σημείο. Αν συμφωνούμε 100% με αυτά που λέγαμε ΔΕΛΤΑ και πούμε ναι μειώνονται οι πόροι, αλλά για κάποιες περιφέρειες έρχονται άλλα έγγραφα. Και κάποιες περιφέρειες και περιοχές λένε θέλουμε περισσότερα χρήματα, άρα πρέπει ξεχωριστά να μας δώσετε περισσότερα. Και μετά έχετε άλλη περιφέρεια και άλλη χώρα. Πώς να τα πω. Πρέπει να είμαστε λίγο συντηρητικοί νομίζω. Καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι περιφέρειες είναι απομονωμένες, είναι μακρινές και πρέπει να τις στηρίξουμε, αλλά η κατάσταση έχει ως εξή. Όλη η κατάσταση έχει ως εξή. Δεν έχουμε χρήματα, τόσο όσα θα θέλαμε. Και πρέπει κάπως να το λύσουμε με αλληλεγγύη, αλλά δεν μπορούμε να ε, αγνοούμε το γεγονό ότι αν βοηθήσουμε κάποιε περιφέρειες μετά θα έρχονται άλλε και θα μα ζητάνε περισσότερα χρήματα. Επαναλαμβάνω αυτές τις προτάσεις ΓΔ Ρέτζι έρχονται, είναι στο δρόμο. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να δούμε πώ θα αντιδράσουμε. Γιατί μιλάμε για πολύ σοβαρέ αλλαγέ ό,τι αφορά του ε, πόρου τα ποσά. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλά προβλήματα για ανταγωνιστικές περιφέρειες, για παράδειγμα. Χρειάζεται αυτή η αύξηση ή όχι. Αν υπάρξει και μείωση των ψώσεων πληρωμών του χρόνου. Προσπαθώ να σας τα εξηγήσω και να τα βάλω σε ένα πλαίσιο τα πράγματα. Αν δείτε την έκθεση απομονωμένη, τι θα πει 0,99 δις, 0,92 δις, ποια είναι η διαφορά. σε πραγματικές τιμές ώστε να είναι ε, λίγο υψηλότερη μέσα. αλλά συγκριτικά είναι υψηλότερη Και αυτό είναι, το, είναι κομμάτι του όλου μηχανισμού. Πρέπει να είμαστε συντηρητικοί. να πούμε ναι κάνουμε αυτό αυτή τη φορά αλλά μετά θα έχουμε 100% προτάσεις από τη ΓΔ Ρέτζι. χωρίς το Connecting Europe είναι πολύ μικρότερο το ποσό στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο από είναι τώρα. Πρέπει να δούμε το πλαίσιο, Ποιε θα είναι οι προτάσεις που θα έρθουν. Αυτέ είναι οι προτάσει. Βέβαια, ουσιαστικά ε, φάσκω και αντιφάσκω λίγο, γιατί άλλα λέω εδώ και άλλα θα πρέπει να πω στα Επιτροπή Ρέτζι. Ε, είναι επικίνδυνο όμω. Έχουμε τα contingent regions, τα competitive regions, remote regions κτλ. Ωραία, μπορούμε να πούμε αύξηση σε όλα, αλλά δεν έχουμε λεφτά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε συντηρητικοί. Και αυτή είναι η πρόταση που έχω να σας κάνω για την όλη συζήτηση. Θα δείτε και στο Κόμπου News τον Απρίλιο του 12 νομίζω πρέπει να εγκριθεί στην Ολομέλεια. Μέχρι τότε θα έχουμε πολλές προτάσεις. και για το 2,5 και για τις ε, περιοχές που είναι στη φάση της μετάβασης και ούτω καθεξής. Έχω τις αμφιβολίες μου πάντως. Δεν πρέπει να απομονώσουμε το ένα από το άλλο αν τα δούμε τα πράγματα διαφορετικά για κάθε περίπτωση, δεν θα μας μείνει φράγκο μετά. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπει κανείς τα πράγματα σφαιρικά και συνοπτικά σε συνεργασία με την Επιτροπή Περίφ που είναι και η αρμόδια επί της ουσίας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν βλέπω να ζητάει κανείς ή καμία το λόγο. Σας επιβεβαιώνω λοιπόν ότι θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης του συναδέλφου 25 και 26 Ιανουαρίου η διορία για την κατάσταση των προβιών την 1η Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 8 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ, τίποτε άλλο, κανένα στα διάφορα. Η any other business, όχι, η συνεδρίαση, θα ξαναειδωθούμε τη Δευτέρα στο Στρασβούργο στα 21 η ώρα. και